Ehm, Καλημέρα συνάδελφοι, συγγνώμη την καθυστέρηση. Ξεκινάμε αυτή τη τελευταία συνεδρίαση των εργασιών μας πριν από τις ε, θερινές διακοπές. Σας ρωτώ αν έχετε αντιρρήσεις, αν έχετε αντιρρήσεις να εγκρίνουμε τα πρακτικά της 8 Ιουνίου. Όπως σας ενημερώσαμε και όπως έχετε και στο χαρτοφύλακα στα πρακτικά, δεν έχετε αντιρρήσεις, όχι, Εγκρίνοντας, σας υπενθυμίζω ότι αυτή η συνεδρίαση μεταδίδεται μέσω web streaming στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου. Και πάμε αμέσως στο σημείο 4, διότι σήμερα έχουμε εισηγητή τον κύριο Γιακολίνα, που ήδη έχει παρουσιάσει το σχέδιο έκθεσης κατά τη διάρκεια της ε, συναντήσεως της 18 Ιουνίου. Ε, σήμερα ξέρουμε ότι έχουν υποβληθεί 392 τροπολογίες, κύριε Γιακολίνο. Για μία ακόμη φορά αυτό δείχνει την προσοχή από πλευράς των συναδέλφων όσον αφορά τις εργασίες αυτής της Επιτροπής παρά κάποιες ε, μικρές εργασίες. Πάντων. Λοιπόν, έχουμε 392 τροπολογίες και αυτή η συζήτηση έχει σαν σκοπό να διευκρινίσει ακόμα καλύτερα τις διάφορες θέσεις των συναδέλφων που παρουσίασαν τις διάφορες τροπολογίες. Θα σας δώσω ένα 20 λεπτό χρόνο αγόρευσης, ούτω ώστε να κάνετε μια παρουσίαση και μετά ε, θα δώσουμε τρία λεπτά στον κάθε συνάδελφο, ξεκινώντας από τους συντονιστές. Λοιπόν, έχετε το λόγο κυρία Γιακολίνο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όπως σωστά υπενθυμίσατε πριν από λίγο και σε αυτή την περίπτωση δόθηκε πολύ μεγάλη προσοχή στην έκθεση που είναι στο τέλος θητείας 392 πράγματι τροπολογίες έχουν υποβληθεί οι από αυτές που κατετέθησαν όσον αφορά την έκθεση, στο, τη συνδιάμεση έκθεση αυτή η μεγάλη συμμετοχή και οι γραπτές συμμετοχές είναι αντιστρόφως ανάλογοι ε, στην συμμετοχή στις συνεδριάσεις που όπως υπενθυμίσατε, πώς να σας πω, ε, είναι αξιολογούνται από όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Υπενθυμίζω ότι η έκθεση αυτή ενδιάμεση χαρακτηρίστηκε από 77 συμβαστικές τροπολογίες επεδείχθη μεγάλη διθεσιμότητα ε, συνεργασίας με τις ομάδες και ενδιάμεση έκθεση μετά αποτέλεσε αντικείμενο έγκρισης ε, για να και και στο, στη συνομιλία του Ιουνίου στο Στασβούργο. Ευχαριστώ τη Γραμματεία, τους διάφορους συναδέλφους επικεφαλής ομάδων, τους συντονιστές και ευχαριστώ και όλους εκείνους ε, που στο Προεδρείο κατέβαναν προσπάθειες για να προωθηθεί αυτή η δραστηριότητα που έχει μια υπεραξία ε, και είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Πάμε λοιπόν στις ε, τροπολογίες, οι τροπολογίες που υπευλήθησαν, που κατετέθησαν σε κάποιες περιπτώσεις αποτελούν μια συνεισφορά αξιέπονη, πολύτιμη βελτιώνουν ένα προϊόν που θεωρούμε ότι μπορεί να είναι πιστικό και χρήσιμο για τις αστυνομικές δυνάμεις, τις ερευνητικές δυνάμεις, τις δικαστικές αρχές, αλλά και για τα κράτη-μέλη. Σε κάποιες περιπτώσεις πιθανότατα πρόκειται περί τροπολογιών που επαναλαμβάνονται ή αλληλοκαλύπτονται και δεν προσθέτουν τίποτα συγκεκριμένο στις εργασίες που έχουν διεξαχθεί μέχρι τώρα. Βεβαίως εγώ θα είμαι διαθέσιμος μαζί με τις άλλες ομάδες να εξετάσουμε συμβαστικές τροπολογίες ούτως ώστε να δώσουμε κάποια ουσία ε, στις εργασίες μας. Λοιπόν, για να συνοψίσουμε τις εργασίες και να δώσουμε ουσία θέλω να αναφέρω και το εξή. Η έκθεση αυτή ενδιάμεση είναι κάτι αξιέπαινο και χαρακτηρίζεται από εύρος μεγάλο εύρος κάλυψης. Θεωρήσαμε ότι στην τελική έκθεση θα έπρεπε να μειώσουμε και να εξορθολογήσουμε το περιεχόμενο ε, σε ένα πραγματικό κατάλογο προτεραιότητων για την αντιμετώπιση της διαφθοράς του οργανωμένου εγκλήματος και της, ε, του ξεπλήματος χρήματος. Ε, έχουμε προβλέψει και στο, στην τελική έκθεση να κάνουμε μια πρόβλεψη να, να, να αναφέρουμε διάφορα στοιχεία που θα συμπεριθούν στο τελικό κείμενο όπως το κείμενο που είχαμε συμφωνήσει στην ενδιάμεση έκθεση στο Στρασβούργο. Λοιπόν, πάμε πιο συγκεκριμένα σε κάποια θέματα. Το εμπόριο ανθρώπων, συζητήσαμε κάποιες τροπολογίες που συμπεριλήφθησαν στις συμβαστικές προτάσεις. Άλλες τροπολογίες δεν συμπεριλήφθησαν, επανεπιβλήθησαν. Οι συνάδελφοι Σόντεργαρ και Ντεγιόγκ προσπάθησαν να ετοιμάσουν τελικό κατάλογο των διαφόρων προτεραιοτήτων. Πρόκειται περί προσπαθίας που κατεβλήθη ε, και εγώ ίδιος έπρεπε να επανυποβάλλω με την υποστήριξη της γραμματείας κάποιες ε, τροπολογίες διαγράφοντας κάποια τμήματα του κειμένου ε, αναφέροντας αυτά σε μία αλλού στο κείμενο κείμενο το οποίο ουσιαστικά καθορίστηκε λάβαμε υπόψη κάποιες προτάσεις του ECR και άλλες προτάσεις που σίγουρα θα λάβουμε δεόντως υπόψη ε, ε, λαμβάνω υπόψη ότι η Μεγάλη Βρετανία αυτές τις ημέρες κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες όσον αφορά την, το ένταλμα σύλληψης, το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και την δικαστική συνεργασία. Δηλαδή κινείται προς μια κατεύθυνση που θέλαμε να ακολουθηθεί, δηλαδή της δικαστικής συνεργασίας και αστυνομική συνεργασία με βάση την εμπιστοσύνη μεταξύ κρατών μελών. Και πρόσφατα οι εισαγγελείς που είπαμε ε, έδειξαν στις χώρες τους ότι ήταν στην πρώτη γραμμή της αντιπαράθεσης με το οργανωμένο έγκλημα και όλα αυτά δείχνουν ότι οι ακροάσεις που έλαβαν χώρα ε, συμπεριέλαβαν σημαντικές προσωπικότητες, συμμετοχή σημαντικών προσωπικότητων που ε, ξέρουν πολύ καλά το οργανωμένο έγκλημα και μπορούν να αντιφταχθούν στεναρά έναντι των εγκληματικών οργανώσεων. Η κυρία Αλφάνο και η κυρία Φαγιών αναφέρθηκαν στα χαρτονομίσματα των 200 και 500 ευρώ προβλέποντας δυνατότητα ανιχνευσιμότητας. Το λαμβάνω αυτό υπόψη και η κυρία Καρόν αναφέρθηκε στην οικολογική μαφία ε, και άλλα κείμενα που αφορούσαν ε, διάφορες συμμορίες, την αποποινικοποίηση ε, όπως και το αδίκημα της δυσφήμισης. Η κυρία Γκόμες αναφέρθηκε στα διάφορα στις κατασχεθήσεις περιουσίες, ε, νέους πόρους για τους διάφορους οργανισμούς, ε, η Βερονίκ Μαθιέ, ο Νιούτον Ντάν υπέβαλαν σχετικές τροπολογίες ε, και άλλοι. Επίσης, τροπολογία που αφορούσε τον ρόλο των διαφόρων οργανώσεων και που πρέπει να προβλέπεται, που θα προβλεφτεί αυτή η μερίδα όπου θα τιμούνται, θα, γίνεται, θα θυμόμαστε τα θύματα της μαφίας. Δεν ξέρουμε, θα μπορούσαμε να έχουμε κάποια άλλη μερομή θα βρούμε και να γίνεται αυτή η τελετή σε επίπεδο των κρατών μελών. Αυτό είναι κάτι που θα το διευκρινίσουμε τις επόμενες ημέρες. Κλείνοντας, κυρία Πρόεδρε, πολύ πιο σύντομα από το χρόνο που είχατε τη γενοδορία να μου διαθέσετε, αναφερόμενος ε, στην τελευταία σελίδα μια τροπολογία μου της 387 δεν την διαβάζω για λόγους χρόνου αλλά έχω εκεί συμπυκνώσει όλα τα στοιχεία τα ουσιαστικά προτεραιότητες, στόχους της προσπαθίας που καταβάλουμε όλοι ορισμός του οργανωμένου εγκλήματος, οργανώσεις ε, τύπου μαφίας, ε, ε, φορολογική παράδειση στην Ευρώπη, τα παράνομα έσοδα του εγκλήματος, η οργάνωση, η χειραγώγηση αθλητικών εκδηλώσεων, αντιμετώπιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενίσχυση των διαφόρων συμφωνιών συνεργασίας, κατάσχεση, αμοιβαία αναγνώριση των ποινών. Ε, λοιπόν, να μην μπορέσουμε να μετέχουν σε δημόσιου διαγωνισμούς οι διάφορε εταιρείε που καταδικαστεί η συμμετοχή σε αυτέ τι δραστηριότητε και την ευθύνη του πολιτικού κόσμου και κάποιες αναφορές όσον αφορά το έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Πάνω εδώ και 15 μήνες ξεκίνησα, νομίζω 2012 ξεκινήσαμε, τον Ιούλιο του Ξεκινήσαμε, είμαστε το 2013, τον Ιούλιο του 2013, 15 μήνες εργαστήκαμε σκληρά, συζητούμε διάφορα ζητήματα και θέματα. Τώρα είναι πολύ γνωστά αυτά τα θέματα, αποτελούν τμήμα της κληρονομιάς μας αν θέλετε. Θα έλεγα λοιπόν ότι σε αυτή τη φάση, εκτός ε, αν υπάρξει και ε, ε, άλλη, συνάντηση να συζητήσουμε τις τροπολογίες και τις συμβαστικές τροπολογίες, Κάτι που ελπίζω να το καταφέρουμε το κάνουμε άλλη μια συνεδρίαση προβλέπεται να γίνει την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και στις 17 θα γίνει ψηφοφορία όσον αφορά την τελική έκθεση της Επιτροπής μας και σε αυτό το στάδιο πιστεύω ότι αυτό είναι το πλαίσιο αναφοράς, το γενικό πλαίσιο αναφοράς που μπορούσα να προσφέρω ε, για να έχετε υπόψη σας υπενθυμίζοντας όλους μας ότι όσον αφορά αυτό το θέμα θα ήταν ευκταίο να έχουμε στο τέλος μια ψηφοφορία που θα χαρακτηρίζεται από την ομοφωνία των απόψεων. Λοιπόν, για να εγκριθεί, ότι εγκρίθηκε λοιπόν η ενδιάμεση έκθεση και αυτό γραμμίζεται με τις επιθυμίες του συγκητού που έκανε ό,τι ήταν δυνατόν ακόμα και το ανέφικτο προσπάθησε για να υπάρχει ισορροπημένος ορισμός, σωστή προσέγγιση όσον αφορά την έκθεση που είναι ιδιαίτερα σημαντική αυτή η έκθεση για όλη την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση θα δώσω να καλωσορίσω τον συνάδελφο Ρούσα Τόματζιτ. Ρόζα Τόματζιτς, τη Ρόζα Τόματζιτς που εκπροσωπεί την Κροατία που έχει ενταχθεί πρόσφατα στην Κροατία. Καλωσορίζουμε την συνάδελφο και εκπροσωπεί το ECR. Καλώς. Ξεκινάμε τη συζήτηση. Η συνάδελφος Βερονίκ Ματιό έχει το λόγο για ένα τρίλεπτο. Έχεις τρία λεπτά στη διάθεσή σου, Βερονίκα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν θα χρειαστώ τόσο χρόνο. Θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή μας για την προσπάθεια την οποία έχει ήδη κάνει στα πλαίσια αυτής της τελικής μορφής της έκθεσης του. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που κατέθεσαν τροπολογίες. 392 τροπολογίες αποδεικνύουν το ενδιαφέρον των συναδέλφων στις εργασίες μας. και γενικότερα για το ενδιαφέρον τους ε, και το ενδιαφέρον των μιλών της Επιτροπής μας. Θυμίζω ότι επιθυμία όλων των συναδέλφων και των συναδέλφων της Ολομέλειας ήταν να προχωρήσουν προς την κατεύθυνση αυτή. Έχουμε μπροστά μας την τελική έκθεση λοιπόν, τροπολογημένη στην αρχική φάση ε, στα μέσα της εντολής είχαμε 700 τόσες τροπολογίες που δείχνουν τις ανησυχίες των συναδέλφων στα πλαίσια της καταπολέμησης της εγκληματικότητας, ε, του ξεπλήματος ε, και της διαφθοράς, της καταπολέμησης της διαφθοράς. Ο εισηγητής ασχολείται με όλα αυτά με συστηματικό τρόπο, με την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, με τη σωματεμπορία, με τις μαφιόζικες οργανώσεις, με τα χαρτονομίσματα των 200 και των 500 ευρώ, ε, γενικά συμφωνώ πως ε, και ο ίδιος ο εισηγητής το Σεπτέμβριο να καταλήξουμε σε συμβιβαστικές τροπολογίες και να καταλήξουμε σε μια πολιτική η οποία ε, θα καλύψει τις ανησυχίες μας για αυτή τη μάστιγα. Ε, συζήτησα και με τη Λιθουανική Προεδρία τη συγκεκριμένη έκθεση. Αναφερθήκαμε στις ανησυχίες και τις προτεραιότητες της Λιθουανικής Προεδρίας και η έκθεση αυτή ε, περιλαμβάνεται στις προτεραιότητες αυτές, στις προτεραιότητες του Υπουργού Εσωτερικών με τον οποίο μπόρεσα ήδη να συζητήσω για τις ανησυχίες που έχουμε. Θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας λοιπόν στην οργανωμένη αυτή εγκληματικότητα, μορφή εγκληματικότητας στα πλαίσια της Λιθουανικής Προεδρίας. Ευχαριστώ κυρία Ματιέ. Φαγιόν τρία λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Σαλβατόρα για την εκθέση αυτή και για τη δουλειά που έχει κάνει και να ευχαριστήσω και τους κοινωνισηγητές, συντονιστές και λοιπούς. Ελπίζω οι τροπολογίες μας να βελτιώσουν το κείμενο και θα ήθελα πραγματικά να ληφθεί υπόψη το κείμενο αυτό από τις κυβερνήσεις το φθινόπωρο. Η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς ε, γίνεται ένα το ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πρόβλημα. Είναι σαφές πως δεν είμαστε αποτελεσματικοί στην καταπολέμηση αυτής της μάστιγας. Ε, η ομάδα μας έχει πολλές απολογίες τώρα. Να αφαιρεθώ σημαντικότερες. Πρώτα απ' όλα εμπορία ανθρώπων. Ένα ζήτημα που πλήττει όλα τα κράτη-μέλη. Είτε ως χώρες διέλευσης, είτε ως χώρες τελικού προορισμού. Και δεν έχουν κυρώσει τα κράτη-μέλη όλες τις διεθνείς συμφωνίες ακόμα για να καταπολεμηθεί σωστά το φαινόμενο. Γι' αυτό πρέπει ξανά και ξανά να επισημάνουμε το ζήτημα αυτό. Γιατί τα, τα θύματα τελικά ε, απομένουν στο έρμεο των διακινητών. Δεν έχουν έγγραφα, ζουν με φόβο και πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Οι συμβαστικές μας προτάσεις νομίζω θα μπορέσουν να ικανοποιήσουν τους πάντες εδώ πέρα. Τώρα, για τους μετανάστες θα ήθελα να πω πως στις τροπολογίες μας λέμε πως ε, πολλά κέντρα κράτησης δεν ε, μεταχειρίζονται ε, σωστά τους ανθρώπους αυτούς. Επίσης μιλήσατε για τα 200 ευρώ και τα 500 ευρώ. Να πω πως στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ συντάσσουμε μια έκθεση που στόχο έχει την καταπολέμηση των ε, περιστατικών ε, ξεπλήματος χρήματος και μέσω επίσης της εκτύπωσης πλαστών ε, χαρτονομισμάτων. Οι ελάχιστες λοιπόν αρμονισμένες κυρώσεις είναι νομίζω μια πρόταση όταν μιλάμε για τουλάχιστον 10.000 ευρώ να έχουμε τουλάχιστον φυλάξει 6 μηνών. Ο κύριος Γιακολίνο και εγώ πάντα επισημέναμε πως ε, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη εγκληματικότητα στο τομέα της γεωργίας και των τροφίμων. Ειδικά στα κράτη-μέλη όπου που δίνουν ιδιαίτερη σημασία στο, στα ποιοτικά τρόφιμα. Τώρα για το τζόγο και τα καζίνο πρέπει να διαγραφεί το κομμάτι που μιλάμε για τον νόμιμο τζόγο γιατί ο, ο τζόγος δεν είναι νόμιμος σε όλα τα κράτη-μέλη. Για τα νόμιμα και τα, για τζόγο τώρα και τα νομικά συστήματα είναι σαφές πως ε, τα νομικά συστήματα δεν είναι αρκετά αποτελεσματικά και δεν τα εμπιστεύεται ο πληθυσμός. Γι' αυτό πρέπει να ξαναλέμε πως η αποτελεσματική δικαιοσύνη έχει μεγάλη σημασία και επίσης τα δικαστήρια δεν πρέπει μεροληπτούν. Και άρα πρέπει να είναι ανεξάρτητοι και οι δικαστές. Αυτά είναι σημαντικά για μένα και την ομάδα μου. Ελπίζω να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποιους συμβιβασμούς και μετά το Σεπτέμβρη να έχουμε ποιοτικές προτάσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Φαγιό. Ο Νιούτον ήταν τρία λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι σημαντική στιγμή. Έχουμε δουλέψει πολύ τους τελευταίους 12 μήνες, έχουμε συλλέξει πάρα πολλές πληροφορίες και τώρα πρέπει να δώσουμε μια καλή έκθεση για να μην πάνε χαμένα αυτά που έγιναν. Είναι δύσκολη στιγμή, κρίσιμη. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό πράγμα το οποίο μπορούμε να κάνουμε σαν Επιτροπή είναι να βεβαιωθούμε ότι όταν τελειώσουμε και πρέπει να τελειώσουμε τον Οκτώβριο να μην πάει χαμένη η δουλειά μας. Να αφήσουμε ένα ίχνος σε πάση περιπτώσει για το τι θα κάνουν οι μελλοντικοί βουλευτές. Τι θα κάνει το νέο κοινοβούλιο θα δημιουργήσει και αυτό μια υποεπιτροπή, μια επιτροπή θα πει ότι καλά ήτανε αλλά τελειώσαμε το 13 με όλα αυτά. Θα πρέπει να αποφασίσουμε λοιπόν από κοινού για να δούμε ποιο θα είναι το επόμενο βήμα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για το τι θα πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί του ζητάμε πάρα πολλά πράγματα. Θα υπάρξει νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή του χρόνου και θέλουμε και από αυτού να μάθουμε κάποια πράγματα πώς το Κοινοβούλιο θα ελέγχει τις εργασίες τους και πώς θα κάνουν αυτά τα οποία το άμεσα εκλεγμένο Κοινοβούλιο του ζητά. Λοιπόν, ε, αυτό είναι το θέμα, τι θα γίνει στο μέλλον και πώς επίσης τα κράτη-μέλη συμπεριφέρονται, όπως ε, είπε και η κυρία Φαγιών, Η ιδέα του να μην επικυρώνουν τις προτάσεις αυτές στα κράτη-μέλη είναι απίστευτη και δεν πρέπει να το καταπιούμε αυτό. Πολλά μένει να γίνουν λοιπόν αυτή τη στιγμή κλείσει η Επιτροπή μας. Μου φαίνεται επίσης ότι έχουν βγει και άλλα πολύ σημαντικά θέματα από τις προσπάθειες που κάνουμε, όπως η αποτυχία των κρατών μελών να εργαστούν, να συνεργαστούν αποτελεσματικά μεταξύ τους, για λόγους ιστορικούς, για λόγους διαφορετικών γλωσσών, συστημάτων, έλλειψης εμπιστοσύνης, και γι' αυτό αυτό που πρέπει κυρίως να συστήσουμε είναι να υπάρχει σωστή διμερή συνεργασία. Οι εγκληματίε είναι πάρα πολύ καλοί όταν δραστηριοποιούνται διαμεθοριακά και τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να συνεργαστούν αποτελεσματικά αυτή είναι τομεί που πρέπει να καλυφθούν λοιπόν. Όντας μέλος και της αντιπροσωπείας προς τη Ουάσιγκτον θα πρέπει να προχωρήσουμε προς μια ομοσπονδιακού τύπου αστυνομία στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε άμεσα βέβαια, απαιτούνται πολλά ενδιάμεσα βήματα. Πρέπει να βοηθήσουμε την Ευρωπόλ να αναπτυχθεί, να μην έχει μόνο την δυνατότητα συλλογής πληροφοριών και με περιορισμένο τρόπο όπως σήμερα, αλλά να βγει στους δρόμους η Ευρωπόλ, να συλλέγει στοιχεία επιτόπου. Και είναι πολύ δύσκολο να έχει κανείς βέβαια αξιόπιστες στατιστικές, αλλά είναι σαφές ότι ε, ε, δεν πρέπει ε, να ξεχνάμε ότι πάρα πολλά είδη που εισέρχονται όχι μόνο από την Κίνα στην Ευρώπη αλλά από όλο τον κόσμο είναι ε, παραποιημένα, είναι ψευδεπίγραφα και αυτό καταστρέφει χιλιάδες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη και αν θέλουμε να ανακτήσουμε τις θέσεις αυτές και να αυξήσουμε τα κέρδη θα βγούμε και από την οικονομική ύφεση, αυτό να μην το αγνοούμε. Ε, όσοι από εμά πήγαμε στη Νέα Υόρκη είδαμε κάτι το οποίο μας επηρέασε αρνητικά. Είδαμε ότι ένας πολύ μικρός αριθμός ε, από τα εμπορευματοκιβώτια που εισέρχονται στο λιμένα ελέγχονται πραγματικά. Ο αστυνομικός υπεύθυνος του λιμένου της Νέας Υόρκης μας είπε ότι ελέγχουν μόνο το 5% αν και ήξερε ότι και τα υπόλοιπα μπορεί να περιελάμβαναν παραποιημένα προϊόντα, κοκαίνη και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Ε, στην Ανβέρσα σαν παράδειγμα εμείς ελέγχουμε το 3% των εμπορευματοκιβωτίων. Το 97% αυτών που εισέρχονται στην Ευρώπη λοιπόν δεν ελέγχονται καθόλου. Υπάρχει τεράστιος χώρος για κοκαίνη, για ψευδεπίγραφα κτλ. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε ορισμένες συστάσεις για το τι ε, πρέπει να κάνουμε στα πλαίσια της αποτυχίας μας να ελέγξουμε τα εμπορευματοκιβώτια που εισάγονται στην Ευρώπη. Και το θέμα της ε, ε, διαμήρασης και κατανομής των δεδομένων και των πληροφοριών. Ο, ο Δήμαρχος Τζουλιάνη στη Νέα Υόρκη πέτυχε με την πολιτική της μηδενικής ανοχής συνδέοντας τις ε, τράπεζες δεδομένων των αστυνομικών δυνάμεων στην πολιτεία. Και ε, τα κράτη-μέλη αν δεν θέλουν να συνεργάζονται στον τομέα αυτό προφανώς ε, δεν θα προχωρήσουμε. Απαιτούνται επίσης και κοινέ πρακτικές σε σχέση με τις καταδίκες, σε σχέση με τις Use the σχέσεις και τα λοιπά. Εδώ έχουμε κάποια αδυναμία γιατί υπάρχουν διαφορές στα κράτη-μέλη. Και πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουμε και την αναπτυσσόμενη δραστηριότητα της εγκληματικότητας στο διαδίκτυο. Απαιτείται και διαφάνεια βέβαια, γιατί ακούσαμε από πολλούς εμπειρογνώμονες ότι η διαφάνεια είναι ε, καθοριστική για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Δεν μπορεί κανείς να είναι διεφθαρμένος και να ε, κάνει κατασκρίσεις εις βάρος του δημοσίου αν υπάρχει διαφάνεια. Ε, γι' αυτό λοιπόν η μελλοντική κληρονομία της Επιτροπής μας θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη. Κοιτάξτε, έχω ίσως ξεπεράσει και το χρόνο μου. Ευχαριστώ που με ανέχεστε. Χτες η Βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα opt-out από τα θέματα εσωτερικών υποθέσεων δικαστικών και αστυνομικών δραστηριοτήτων. Αυτό είναι πραγματικά απέσιο και ηλίθιο. Είναι μια μεγάλη ανοησία αυτή που έκανε η Βετανική κυβέρνηση, ελπίζω να ακουστεί μέσα από το διαδίκτυο σε όλους. Συμβιβαστικά με τους φιλελευθέρους ε, που είπαμε ε, ότι δεν έπρεπε να το κάνουμε, οι συντηρητικοί είπαν θα το κάνουμε, λόγω πραγματικά της ιδιαίτερα αντιευρωπαϊκής συντηρητικής και ακροδεξιάς αντίληψης των συντηρητικών. Αλλά αυτό που δεν υπόθηκε χθε από τη Βρετανική κυβέρνηση και πρέπει να ακουστεί και αυτό από το διαδίκτυο, αυτό το οποίο δεν εξηγήθηκε από την κυβέρνηση γιατί τους ενοχλεί, είναι ότι το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να κάνει ένα opt-out πρώτα από όλα τα άλλα και πρέπει να αναδιαπραγματευτεί δηλαδή ε, την συμμετοχή τους στα 35 μέσα τα οποία υποτίθεται εξακολουθεί να θέλει να χρησιμοποιεί. Αυτό σημαίνει ότι μετά από το βρετανικό opt-out για μήνες ολόκληρους θα είμαστε απροστάτευτοι απέναντι στην διεθνή εγκληματικότητα. Γιατί, ε, δεν, ε, θα, θα, γιατί θα μεσολαβήσει χρόνος έτσι ώστε να τεθούν σε λειτουργία τα 35 μέτρα τα οποία θέλει να θέσει ε, σε ισχύ η Βρετανική κυβέρνηση. Λοιπόν, αρνείται τη συνεργασία με την Ευρώπη και με όλο τον κόσμο ουσιαστικά για πάρα πολλούς μήνες. Ε, ξέρετε ότι θα έχουμε του χρόνου και νέο κοινοβούλιο και νέα επιτροπή. Είναι τόσο ανεύθυνη η στάση της Βρετανικής κυβέρνησης και η Βρετανή συντηρητική. Και λυπάμαι που ε, που είναι ένας ε, πραγματικά λογικός συντηρητικός έφυγε από την επιτροπή μας. Λοιπόν πρέπει να αφήσουμε πράγματα όταν σταματήσουμε να δουλεύουμε. Παρακαλώ να κλείσετε λέει η Πρόεδρος πρέπει να καταλήξουμε σε σωστές συμβιβαστικές και να αφήσουμε μια χρήσιμη κληρονομιά για το μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίως που εκφράσατε τις ανησυχίες για τη χώρα σου. Θα δώσω το χρόνο τώρα στον συνάδελφο ε, Μπορσελίνο. Στη συνάδελφο Μπορσελίνο. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω και εγώ ευχαριστώντας την Επιτροπή Ίντερ, ευχαριστώ την Πρόεδρο όλες ιδιαίτερος, ευχαριστώ τη Γραμματεία και όλους τους συναδέλφους βεβαίως και τον εισηγητή, τον κύριο Γιακολίνο και όλους εκείνους που εργάστηκαν με προσοχή και με ενθουσιασμό επεξεργαζόμενοι το θέμα αυτό. Ήδη η καινοτομία της αντιμετώπισης του θέματος πιστεύω ότι είναι κάτι σημαντικό και ο αριθμός των τροπολογιών που είναι πολύ μεγάλος, που υπευλήθησαν, είναι σημάδι μεγάλης προσοχής. Που δεν τονίζεται βέβαια από τη συμμετοχή, που δυστυχώς είναι πάντα ρεή, αλλά υπάρχει και το πρόβλημα ότι ταυτόχρονα υπάρχουν και άλλες ε, εργασίες σημαντικές που διεξάγονται. Και δυστυχώς αυτό ε, είναι εις βάρος των εργασιών μας. Πιστεύω όμως ότι αν κάνουμε ένα απολογισμό πρέπει να πούμε ότι πραγματικά η προσοχή των θεμάτων που συζητήθηκαν στην Επιτροπή όσο αυτά τα θέματα αυτά ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Ήταν ε, σημαντικό αυτό που έγινε και καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα με καινοτόμα στοιχεία. Να μην εξετάσουμε το θέμα με γνωστά επιχειρήματα που θα επικαιροποιούνται, αλλά καινοτόμα προσέγγιση ακολουθήσαμε. Και νομίζω ότι αυτό είναι το στοιχείο το σημαντικότερο οι τροπολογίες που έχουν υποβληθεί, όπως έλεγε ο κ. Γιακολίνο, σε κάποιες περιπτώσεις υπογραμμίζουν και εμβαθύνουν σε θέματα που ήδη αναφέρονται στην έκθεση. Υπάρχουν όμως και κάποιες τροπολογίες όπως η οικολογική μαφία που έχουν ε, καλυφθεί κάπως και έπρεπε να υπογραμμιστεί. Άρα αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Αυτό το ζήτημα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Εξάλλου είναι κάτι που ενδιαφέρει όλη την Ευρώπη και όχι μόνο κάποιες χώρες. Το ίδιο ισχύει και για το εμπόριο ανθρώπων. Συζητήθηκε και συζητείται και αναφέρεται στην έκθεση, αλλά το να υπογραμμίσουμε κάποια πράγματα και να τα εμβαθύνουμε πιστεύω ότι είναι κάτι που ποτέ δεν αποτελεί πλεονασμό. Και ο κύριος Μωράες ήθελε να υπογραμμίσει την παράνομη μετανάστευση. Πιστεύω ότι είναι κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η λαθρομετανάστευση δεν είναι πάντα παράνομη, θεωρείται παράνομη και πρέπει να δώσουμε προσοχή και στη διπλή δίωδο που χρησιμοποιεί το εμπόριο ανθρώπων. Δηλαδή υπάρχει οικονομικό όφελος για τους εγκληματίες και υπάρχει και άλλη πτυχή, η πτυχή που αφορά τα θύματα αυτά κάθε αυτά. Τροφοδοτείται η, η μαύρη αγορά και τροφοδοτείται επίσης και το κύκλωμα της πορνείας. Στο γεωργικό τομέα αναφέρθηκε Υπάρχουν ε, διάφορες διαδικασίες που αφορούν τα τρόφιμα. Είναι ένα πρόβλημα πάρα πολύ περίπλοκο, σοβαρότατο και κάτι άλλο το οποίο υπεγραμμίστηκε μέσω των τροπολογιών της ομάδας μου. Μέσα στα ε, ευρω... στους εντάσσονται τρία θέματα. Το εμπόριο των αποβλήτων, των έργων τέχνης και των προστατευμένων ειδών. Είναι, ε, θα πρέπει να παριθμηθούν αυτά μέσα στα εγκλήματα. Η ανεχνευσιμότητα των χαρτονομισμάτων αναφέρθηκε. Πρέπει να δοθεί προσοχή και στον, στην ερευνητική δημοσιογραφία. Πρέπει να δοθεί προστασία στην ερευνητική δημοσιογραφία. Όσον αφορά μια διευκρίνηση. Δηλαδή, να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα η απάτη που στρέφεται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Να μην επιβάλλονται μόνο διοικητικές κυρώσεις. Τέλος, όσον αφορά την ημερίδα αυτή της ανάμεσης των θυμάτων, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο να υπάρχει μια ημέρα που να θυμόμαστε τα αθώα θύματα των, του οργανωμένου εγκλήματος και της μαφίας. Στην Ιταλία εδώ και 18 χρόνια, 21 Μαρτίου είχε επιλεχθεί, διότι είχε σημασία ιδιαίτερη. Η πρώτη μέρα της Άνοιξης είναι 21 Μαρτίου, δηλαδή δείχνει ανανέωση, ότι ξεκινάμε από την αρχή, ξαναδημιουργείται εμπιστοσύνη, ακόμα και σε εκείνους που έχουν ζήσει τις εμπειρίες. 21 Μαρτίου ίσως θα μπορούσε να γιορτάσετε αυτό σε διάφορες χώρες, θα μπορούσε να καθοριστεί άλλη ημερομηνία. Αλλά εφόσον υπάρχει από παλιά μία ημέρα και μία ημερομηνία, κατά την άποψή μου θα ήταν σημαντικό μήνυμα να δώσουμε μία συνέχεια στο μήνυμα αυτό, στο πούμε μήνυμα. Θετικό μήνυμα. Να υπογραμμίσω εκ νέου τη σημασία των εργασιών που έλαβαν χώρα. Έπρεπε να αντιμετωπίσουμε υλικό πολύ ογκός, που αυξανόταν ανάμεσα στα χέρια μας, διότι κάθε θέμα ε, συμπαρέσυρε κι άλλο θέμα και γι' αυτό χρειάστηκε να γίνει τόση δουλειά, να δοθεί τόσο προσοχή σε ένα θέμα που ουσιαστικά περιθωριακά εξεταζόταν μέχρι τώρα. Ελπίζω ότι όλη αυτή η προσπάθεια να έχει σημαντικό βάρος στη συνέχεια που θα δοθεί, στην προσοχή που θα δοθεί στα θέματα αυτά. Να μην παραμείνει αυτή η δουλειά μια πρωτοβουλία όμορφη που εσωκλίνεται στον εαυτό της. Ελπίζω και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει πραγματικά να συνεχίσει ακολουθώντας αυτό τον δρόμο που ανοίξαμε. Ευχαριστώ κυρία Μπορσελίνο. Υπάρχει άλλος που θέλει το λόγο. Όχι. Πριν ξαναδώσω το λόγο... Α, ορίστε. Έχετε το λόγο. Ζόμπρο. Ξανά Ζόμπρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και το προσωπικό που προετοίμασαν αυτό το έγγραφο. Να αναφέρω κάποια ζητήματα που ακούστηκαν στη συζήτηση και είναι πολύ σημαντικά. Και ίσως μπορούμε να τα υπογραμμίσουμε στις συμβαστικέ προτάσεις. Αναφέρομαι σε ζητήματα που είναι γνωστά αλλά δεν έχουν ακόμα εφαρμοστεί, δηλαδή την ε, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων ε, που έχουν προκύψει από το οργανωμένο έγκλημα, αλλά επίσης και τα εισοδήματα από παράνομες πράξεις. Αυτό λοιπόν από πλευράς ε, εφαρμογής διαφέρει από χώρα σε χώρα. και είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μέσο όσον αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Αυτό το πρόβλημα το βλέπω και στην Πολωνία. Μέτρα δηλαδή τα οποία ουσιαστικά επιτρέπουν στις αρχές να κατασχέσουν ε, ε, περιουσιακά στοιχεία τα οποία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο συνδέονται με δραστηριότητες οργανωμένου εγκλήματος. Από όσο ξέρω υπάρχουν ακόμα τέτοια εμπόδια σε τη μελη οπότε θεωρώ πως η εισαγωγή τέτοιων κανονισμών είναι πάρα πολύ σημαντική. Κάτι άλλο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω είναι η σημασία κοινών ε, ερευνητικών ομάδων στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω πως η φύση ε, του οργανωμένου κλίματος ε, καθιστά αυτό το ζήτημα απολύτως απαραίτητο. και οπωσδήποτε θα συνεισφέρει στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Ως υπουργό Δικαιοσύνης ε, και εισαγγελέα είχα ασχοληθεί με τέτοιες ε, έρευνες στην Πολωνία και στην Ιταλία και Γνωρίζω τα ωφέλη της ε, καλής συνεργασίας, αλλά βεβαίως είχα να αντιμετωπίζω και την έλλειψη νομοθεσίας που θα επέτρεπε την δημιουργία τέτοιων κοινών ερευνητικών ομάδων. Ελπίζω λοιπόν να εισαχθούν ευρύτατες αλλαγές για να μπορούν να δημιουργηθούν τέτοιε ομάδες όπου αυτό είναι απαραίτητο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφε Ζόμπρο. Συνάδελφε Σμίτ, έχετε το λόγο. Σύντομα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συγκεκριτή και να τονίσω αυτό το οποίο είπε ο Μπιλ Νιούτονταν. Και για την Βρετανία βεβαίω. Είναι καταστροφή αυτό το opt-out, αλλά πάντων. Για τη συνεργασία. Τώρα, θεωρώ πως πρέπει να κάνουμε περισσότερα και το κείμενο της έκθεσης ε, κάπως ε, ασθενές έπρεπε να είναι αυστηρότερο. Αλλιώς, κατά την άποψή μου, δεν θα λύσουμε τα προβλήματα εάν ε, δεν δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή αστυνομία ή όπως θέλει κανείς να το πει. Να σας δώσω ένα πρακτικό παράδειγμα. Γίνεται εμπορία ανθρώπων ε, στην έρημο του Σινά. Ε, ξέρουμε τι γίνεται στην Αίγυπτο. Στην Ερυθρέα, παραδείγματος χάρη. 4.000 άνθρωποι κάθε μήνα φεύγουν από την Ερυθρέα, καταλήγουν στο Σινά. Συγγνώμη, το τηλέφωνο μου. Και απάγονται, βασανίζονται. Και ίσως τους αφαιρούν και όργανα και τα πουλάνε σε άλλες χώρες. υπάρχουν δε λίτρα 30-40 ευρώ που εισπράττονται. Πριν από λίγες εβδομάδες υπήρξε μια δίκη στη Στοκχόλμη. Δύο άνθρωποι που ζούσαν στη Σουηδία κατηγορήθηκαν και καταδικάστηκαν για το θέμα αυτό. Και ξέρουμε πως αυτό συμβαίνει και στην υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά δεν, δεν μπορεί να κάνουν τίποτα. Γιατί ε, το θέμα είναι ακριβώς το θέμα της κοινής ομάδας έρευνας. Γιατί πρέπει η αστυνομία να πει πρέπει να συνεργαστούμε με μια άλλη αστυνομία. Και αυτό είναι περίεργο γιατί γνωρίζουμε πως συμβαίνει κάτι τέτοιο. Τώρα έχουμε την πρώτη απόφαση δικαστηρίου στην Ευρώπη και δεν κάνουμε τίποτα. Αυτό είναι κακό. Αυτό θα ήθελα να τονίσω πως χρειαζόμαστε συνεργασία και ευρωπαϊκή αστυνομία. Ξέρω πως είναι δύσκολο αυτό, ειδικά για τους Βρετανούς και για μας και, και για σας. Αντάξει, ορίστε να. Αλλά εάν είναι να κάνουμε κάτι για το οργανωμένο έγκλημα πρέπει να νομίζω το χρειαζόμαστε αυτό το μέσο και μπορούμε να στηρίξουμε τις τροπολογίες. που ζητάνε επιτάχυνση. Ευχαριστώ, συνάδελφε Βάιλερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Σμιτ. Θα ήθελα να πω κάτι για το θέμα. Εγώ έχω την ελπίδα πως, δεν πότε σήμερα, αύριο, μεθαύριο, θα οριστεί ο πρώτος Ευρωπαίος εισαγγελέα. Γιατί αυτά δεν πρέπει να μένουν μόνο στα χαρτιά. Χρειαζόμαστε μια αρχή με αρμοδιότητες που θα αποκτήσει κάποια ουσία. Αυτό δεν είμαι τόσο απεσιόδοξη. Ελπίζω λοιπόν του χρόνου. Εντάξει τώρα πολύ αργά για την περίπτωση που αναφέρατε, αλλά το αργότερο μετά τις ευρωεκλογέ να ασχοληθούμε σοβαρά με αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ Μπάρμπαρα. Πριν δώσω το λόγο στον συγγητή, να σα υπενθυμίσω κάτι που ήδη αναφέρθηκε 9 Σεπτεμβρίου λοιπόν στο Στρασβούργο λοιπόν θα συζητήσουμε ενδελεχέστερα τις τροπολογίες. Θα είναι έκτακτη συνεδρίαση ΚΡΙΜ και μετά θα λάβει χώρα η ψηφοφορία στην, το απόγευμα της 3ης 17 Σεπτεμβρίου στην ΚΡΙΜ. Εκτός αν γίνουν, υπάρξουν άλλες αλλαγέ, άλλα προβλήματα που ε, εύχομαι να επιληθούν τυχόν προβλήματα αμέσω. Στην παρέμβαση που αναφέρει δική μας επιτροπή τα προβλήματα, στην παρέμβαση λοιπόν που, που έκανε ο κύριος Νιούτον Ντόν, αναφερόμενος στις ανησυχίες του σχετικά με τη δυνατότητα του Ε.Β. Βασίλειου να γίνεται ε, θύμα όλο και περισσότερο του Ενωμένου Βασίλειου των εγκληματικών οργανώσεων, δυστυχώς μπήλει η ανησυχία σου εκ των πραγμάτων υφίσταται, υλοποιήθηκε. Και αναφέρομαι σε αυτό που είπε και ο Σμιτ και η Μπάρμπαρα Βάιλερ. Υπάρχει υποτίμηση από πλευρά πολιτική των κρατών μελών του θέματο. Πολλέ φορέ εδώ αναφέρθηκε λείπει η αποφασιστικότητα και η βούληση από πλευρά κρατών μελών να ακυρώσουν συγκεκριμένε αποφάσει. Όταν αυτή η επιτροπή γεννήθηκε, στόχο είχε όχι μόνο να επεξεργαστεί ένα ενίο κείμενο για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, τη διαφθοράς και του ξεπλήματος χρήματος, αλλά γνωρίζαμε όλοι τέλεια την ανάγκη που υπήρχε να ενισχυθεί και να αξιοποιηθεί η συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και η συνεργασία από πλευρά σε, σε επίπεδο. Τώρα, το ότι αυτή η Επιτροπή αποτέλεσε αξιολόγηση, αξιολόγησης όχι μόνο από διάφορα κράτη-μέλη, αλλά πάνω από όλα από τρίτες χώρες. Η τελευταία μας αποστολή στην Ουάσιγκτον απέδειξε πλήρως αυτό που λέγω, το ενδιαφέρον, τον ενθουσιασμό από πλευράς των αρχών των Ηνωμένων Πολιτειών όσον αφορά τις εργασίες μας ε, και αυτό είναι πρόσφατο γεγονός. Αυτό που πρέπει να αναλυθεί κατά την απόψή μου και να αξιολογηθεί βάθος είναι μέχρι ποιού βαθμού τα κράτη-μέλη και αναφέρομαι εξαιτία του της Ευρωπόλ, μέχρι ποιο βαθμό τα κράτη-μέλη θα κατανοούν ότι χρειάζεται να επενδύσουν. Απόλυτα. σημαίνει πιστεύοντας μέχρι βάθους ότι χρειάζεται επένδυση όσον αφορά την ασφάλεια. Αυτό δεν μπορεί να σημαίνει μόνο καταστολή ή στατικοποίηση. Σημαίνει ελευθερία και δημοκρατία και ασφάλεια για τους πολίτες μας. Πολίτες 28 χωρών. Και αυτό μέχρι τώρα ε, είμαστε μακριά από αυτή την αντίληψη. Και όσο είμαστε μακριά από αυτή την αντίληψη, η δουλειά μας ε, θα είναι να προσπαθεί να δίνει τα στοιχεία επί χάρτου, όλα τα στοιχεία, τα χρήσιμα στοιχεία, ούτω ώστε να μπορούμε να αξιοποιήσουμε, να χρησιμοποιήσουμε και ενισχύσουμε τη συνεργασία. Αλλά όσο θα λείπει αυτή η πολιτική απόφαση, αυτό είναι το αποφασιστικό στοιχείο δυστυχώ, το τελικό στοιχείο, η πολιτική βούληση. Εάν πάμε πίσω ένα χρόνο Σχεδόν κανείς εντός της αιθούσης θα έλεγε τα λόγια που υπόθηκαν σήμερα. Γιατί, διότι εδώ σε ένα χρόνο έγιναν πάρα πολλές ακροάσεις και σε αυτές τις ακροάσεις τα προβλήματα αναφέρθηκαν, εισακούστηκαν, ακούστηκαν διάφοροι πυρογνώμονες, δικαστές, εισαγγελείς, εκπρόσωποι δυνάμεις της, της, της τάξης, δημοσιογράφοι, νομικοί, που παρουσίασαν κάθε πτυχή και έδειξαν ποια είναι η πραγματικότητα, ποιες είναι οι γνώσεις τους. Οπότε καταλάβαμε ότι χρειάζεται να ξεπεράσουμε την ανταλλαγή πληροφοριών, την ανταλλαγή των βελτίστων πρακτικών. Σχετικά με αυτό λοιπόν θέλω να ευχαριστήσω τη γραμματεία, τους συντονιστές, τους συναδέλφους που συμμετείχαν στη συνεδριά της Επιτροπής αυτής. Παρά τις αρχικές ε, προσδοκίες, ε, θεωρήθηκε ότι αυτή η Επιτροπή θα έκανε απλώς μελέτες. Παρά αυτή την άποψη είχαμε το πείσμα των συμμετεχόντων της Επιτροπής. Και έτσι η δουλειά που έγινε καθημερινά έγινε κάτι πραγματικό. Σε βαθμό που εργασίες της Επιτροπής αυτής τώρα θεωρούνται σαν μία από τις προτεραιότητες αυτής της θητείας. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι όταν κανείς έχει γνώση, αντίληψη των πραγματικών προβλημάτων, ε, δεν υπάρχουν ε, προβλήματα ιδεολογικά και πολιτικά. Επικροτώ και ευχαριστώ τους συναδέλφους, διότι αυτή την αίθουσα και συνεδρία των συντονιστών ακόμα ποτέ, μα ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν άκουσα ούτε η διαμάχη, ούτε να ψώνεται φωνή, ούτε να να υπάρχουν προτάσεις πολιτικών ομάδων. Πάντα προσπαθήσαμε να υπάρχει συμφωνία. Ευχαριστώ τον εισηγητή τον κύριο Γιακολίνο, διότι παρά την απόδειξη του ενδιαφέροντος που υπήρξε από πλευρά συναδέλφων, που, δεν είδαμε σε αυτή την αίθουσα ποτέ, παρόλα αυτά που υπέβαλαν τροπολογίες, που είναι κάτι που χαροποιεί αυτό, που σημαίνει ότι υπήρχε ενδιαφέρον όσον αφορά τι εργασίε, ο εισηγητή, πρέπει να πούμε προσπάθησε και βρήκε ε, τρόπο να συνοψίσει τις απόψεις ούτω ώστε 100% να γίνει αποδεκτή αυτή η εργασία. Και είμαι σίγουρη ότι και αυτή τη φορά ε, όσον αφορά τις 392 τροπολογίες θα κάνει την ίδια δουλειά. Σας ευχαριστώ. Δεν ήταν απλή δουλειά και ακόμα δεν είναι. Έχουμε και το τελευταίο στάδιο, το τελευταίο βήμα. Δεν είναι εύκολη δουλειά, όμως σίγουρα αυτό που μέχρι τώρα κάναμε βάζοντας επί χάρτου την προβληματική όπως έλεγε η συνάδελφος Μπορσελίνο, μέσα αυτή την αίθουσα, αυτό το κοινοβούλιο, αντιμετωπίζοντας διάφορα προβλήματα, αυτά δεν είχαν γίνει μέχρι τώρα, δεν υπήρχε η βούληση. Το γεγονός λοιπόν ότι εξετάστηκαν, διευκρινίστηκαν και ότι βρέθηκε το αντίδοτο σε αυτού του είδους ε, τις πτυχές, αυτό είναι σίγουρα κάτι που καθιστά τις εργασίες της Επιτροπής ε, εργασία υψηλού επίπεδου, γι' αυτό ευχαριστώ όλου. ευχαριστώ τη γραμματεία που πάντα έκανε προσπάθεια για να επιλύει τα άλλα προβλήματα. Ευχαριστώ του συντονιστέ και τον εισηγητή για τη δουλειά που έγινε και είμαι σίγουρη ότι θα μείνει στην ιστορία του Κοινοβουλίου αυτή η δουλειά και ελπίζω και εγώ και εύχομαι όπω είπε ο κύριο Νιούτον Ντάν με την ανανέωση, με τη νέα θητεία τον επόμενο Ιούνιο, με την ανανέωση του Κοινοβουλίου ελπίζω να υπάρξει μακρόπνοη ε, προσέγγιση να δούμε ότι αυτό είναι το σημείο άφηξης αλλά είναι η αφετηρία ε, ενός προγράμματος ε, μακρόπνου ευρέως που έχει σαν με έρημνα όχι μόνο την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως αλλά την ασφάλεια και τη δημοκρατία υπέρ των πολιτών μας. Θα δώσω το λόγο αμέσως στον εισηγητή για να δώσει τις απαντήσεις και να εκφραστήσουν αφορά τις σκέψεις που ξέφρασαν οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ συνάδελφε, θα είμαι πολύ σύντομος. Άκουσα με πάρα πολύ μεγάλη ενδιαφέρον τις ομιλίες και τις παρεμβάσεις των συναδέλφων και τη διαθεσιμότητά τους. Οι παρατηρήσεις τους ήταν ιδιαίτερα χρήσιμες. Τους ευχαριστώ και για την εκτίμηση ε, που εξέφασαν απέναντι στην προσπάθειά μας, η οποία όπως ε, θυμίζω ήταν μια ομαδική προσπάθεια του συνόλου των μελών της Επιτροπής απόλυτη προτεραιότητα στα πλαίσια της δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας. Όπως είπε ο Σμιτ, δεν νομίζω ότι το κείμενο είναι ιδιαίτερα ασθενές. Νομίζω ότι είναι αρκετά ενισχυμένο και είμαι πεπισμένος ότι μέσω μιας σωστής αλληλοενημέρωσης και σωστής και στενής συνεργασίας ανάμεσα στις αστυνομικές δυνάμεις, μέσω του συνδυασμού δυνάμεων σε επίπεδο αστυνομικό και ανακριτικό θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε τα οικονομικά και στρατηγικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η στόχη λοιπόν τους οποίους έχουμε θέσει με ξεκάθαρο τρόπο στο κείμενό μας. Τώρα για τη φροντίδα για τους μετανάστες. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Ξέρετε ότι ο Πάπας Φραγκίσκος πήγε στην Ίσο Λαμπεντούσα που είναι τα πραγματικά σύνορα ανάμεσα στον βορρά και στον νότο, ε, νότια της Σικελίας. Στην Ευρώπη και στον κόσμο πολύ σημαντικό σημείο. Έκανε μια πραγματικά ευαίσθητη κίνηση ανάμεσα στους τελευταίους των τελευταίων, τους περιθωριοποιημένους που δεν καλύπτονται από τίποτα. Αλλά το κείμενό μας δεν ασχολείται με αυτό, ασχολείται με το οργανωμένο έγκλημα, με την σωματεμπορία, με το εμπόριο ναρκωτικών και παρόλα αυτά θα πρέπει να δούμε και τα έντονα χαρακτηριστικά τα οποία θα πρέπει να δείχνουν τις προτεραιότητές μας. Επίσης και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα παράνομα κέρδη των, των τυχερών παιχνιδιών. Πολλές φορές ξέρετε ότι με παθολογικό τρόπο ο κόσμος εξακολουθεί να προχωρά σε τέτοιου είδους ε, δραστηριότητες και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και πώς διαφοροποιούνται οι ενέργειες των κρατών μελών στα πλαίσια της αρχής της επικορικότητας. Ε, σε σχέση με αυτά που είπε η κυρία Μπορσελίνο, ε, πράγματι... Τάνια, nella, nella sua, Αναφέρθηκε η κυρία Μπορσελίνο και στις απάτες που μπορεί να γίνονται στα πλαίσια της, ε, των τροφίμων. Ε, μιλήσαμε, εν και για τα χαρτονομίσματα, μιλήσαμε για τα τυχερά παιχνίδια, μιλήσαμε εν μέρη έστω και για τους ε, μετανάστες. Όλοι πιστεύουμε ότι και η υπόθεση του Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα θα μπορέσει να είναι κάτι το χρήσιμο στα πλαίσια της καταπολέμησης των εγκληματικών δραστηριοτήτων και οι κοινέ αστυνομικέ δυνάμεις και ο εισαγγελέα ο Ευρωπαίος μπορεί να είναι ένας στόχος αλλά δεν μπορεί να γίνει κάτι σύντομα ως προς αυτό. Τώρα για τις κοινέ ανακριτικές ομάδες νομίζω αυτό θα είναι ένα καλό και χρήσιμο στάδιο Αναφερθήκατε επίσης στην ερευνητική ε, δημοσιογραφία. Ε, εγώ θα συμφωνήσω και με αυτά που είπε η παρακαθήμενη συνάδελφός μου και για την οικομαφία τη λεγόμενη και για τη μεγάλη σημασία που έχει η δικαστική συνεργασία. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε επίσης ε, και την καταδίκη σε όλα τα κράτη-μέλη της, της ε, δραστηριότητας της αυτοανακύκλωσης των κερδών. Ε, προβλέπονται εδώ διάφορες ποινές ε, οι οποίες θα πρέπει να είναι ανάλογες σε όλα τα κράτη-μέλη. Λοιπόν, έχει μεγάλη σημασία να εξαιρέσουμε από το οικονομικό σύστημα και από τις δημόσιες προμήθειες τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν καταδικαστεί για μαφιόζικες δραστηριότητες σε όλα τα κράτη-μέλη και έτσι θα δώσουμε εγγυήσει για την αξιοπιστία της ευρωπαϊκής αγοράς γιατί οι ε, μη ειλικρινείς και μη ε, νομιμόφρονες επιχειρηματίες θα πρέπει να απομακρύνονται απολύτως από τις ε, διαδικασίες των δημοσίων διαγωνισμών και προμηθειών. Τώρα για το θέμα της υποεπιτροπής το Κοινοβούλιο έχει εκφραστεί πάνω σε αυτό με την ψηφοφορία του. Ήταν σαφής ε, οι προθέσεις του. Αυτό, Πρόεδρε, δεν ε, αναιρεί το ότι πάνω στα συγκεκριμένα θέματα θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια ομάδα εγκαρσίου ε, πολιτικού λόμπι έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την αντιμετώπιση των εγκληματικών αυτών συστημάτων μέχρι το τέλος της εντολής και να επανεκκινήσει η ίδια διαδικασία και με το επόμενο κοινοβούλιο. Συμφωνώ λοιπόν με τους συναδέλφους οι οποίοι πήραν πριν το λόγο. Απαιτείται να υπάρξει ενδυνάμωση και συνέχεια σε αυτήν την ξεκάθαρη επιθυμία την οποία έχει το Κοινοβούλιο λέγοντας ότι η καταπολέμηση των εγκληματικών συστημάτων μπορεί να γίνει μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και για να πετύχει η προσπάθεια αυτή χρειάζεται να συνεισφέρουμε όλοι στον αποκοινού σεβασμό αυτών των αξιών και αρχών. Και κλείνω ότι ε, θα πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας ένα ευέλικτο και σύντομο κείμενο που να ξεκαθαρίζει τις προτεραιότητες με σαφή τρόπο, να διευκρινίζει το τι πρέπει να κάνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να ζητά από το Συμβούλιο να είναι πιο προσεκτικό απέναντι στις δικές μας απαιτήσει και να ζητά από τα κράτη-μέλη να εναρμονίσουν τις ισχύουσες νομοθετικές διαδικασίες ε, σαν παράδειγμα στα σχέση για την αναγνώριση μιας οργάνωσης με χαρακτηριστικά μαφίας όπως έχει πάρει αποφάσεις η Ιταλική κυβέρνηση. Πρέπει λοιπόν μέσω κοινών ε, επιπέδων και αρχών ε, να προσπαθήσουμε να πετύχουμε αποτελέσματα που θα διασφαλίσουν τους Ευρωπαίους πολίτες ε, θα δώσουν χώρο στην πραγματική και τίμια οικονομική δραστηριότητα και θα καταδικάζονται οι ενέργειες οι οποίες είναι παράνομος. Λοιπόν, κλείνω ευχαριστώντας για μια ακόμη φορά όλους τους συναδέλφους οι οποίοι πήραν ε, το λόγο και μέρος. Ε, θυμίζω ότι στις 9 και στις 17 Σεπτεμβρίου λοιπόν θα τα συζητήσουμε αυτά για να καταλήξουμε στις συμβιβαστικές και θα φτάσουμε στην Ολομέλεια τον Νοέμβριο. Η προσπάθεια ήταν δύσκολη, κουραστική, αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι όλοι μπορεί να μείνουμε ικανοποιημένοι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λοιπόν, 9 και 17 Σεπτεμβρίου για την τελική ψηφοφορία σε επίπεδο Επιτροπής. Τώρα θα ήθελα να καλωσορίσω εξ ονόματος της Επιτροπής μας τον κύριο Μισελ Λεβί από το Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ, καθηγητής εγκληματολογίας. Θα μας παρουσιάσει τα προκαταρκτικά αποτελέσματα σχετικά με το κόστος, το πραγματικό κόστος της, του οργανωμένου εγκλήματος. Θα δώσω πρώτο το λόγο για 20 λεπτά λοιπόν στον εισηγητή και αμέσως μετά θα υπάρξει χώρο συζήτησης για τρία λεπτά για κάθε μέλος, το οποίο θα ζητήσει το λόγο. morning, uh, everyone. Micro. Microphone. Okay. Uh, Good morning, everyone. Um, I'm glad that I was able to opt in to this. Καλημέρα. Εγώ χάρηκα που έκανα opt-in στο συγκεκριμένο τέτοιο. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ήρθα σήμερα το πρωί. Ήθελα να κάνω κάποιες αρχικές παρατηρήσεις τώρα για το έργο της Επιτροπής. Θυμάμαι εδώ πέρα το σχόλιο του Βρετανού κομικού Σπαϊκ Milligan πως είμαστε όλοι στο άδειο. Καθαρτήριο θα έλεγε κανείς. Αλλά χαίρομαι που μπορώ να σας μιλήσω για την πολύ προκαταρκτική έκθεση ε, ε, που μπορώ σήμερα να σα παρουσιάσω για τον οικονομικό αντίκτυπο του οργανωμένου εγκλήματο στην Ένωση και στον Ηνωμένο Βασίλειο βεβαίω. Υπάρχει... Υπάρχει μια αγγλική έκφραση που λέει ας ξεκινήσουμε πρώτα από τα του οίκου μας και αυτό το οποίο προσπάθησα να κάνω εγώ και οι συναδελφοί μου είναι και θα είναι βεβαίως πιο εμφανές στην ε, τελική έκδοση είναι να προσπαθήσουμε να δούμε τι μπορεί να γίνει με το έργο αυτό έτσι ώστε εσείς και οι αναγνώστες ε, να αποκτήσετε μια σαφέστερη ιδέα από τη συνήθως για το κόστος του οργανωμένου εγκλήματος. Ένα θέμα το οποίο βεβαίως δεν είναι πάρα πολύ αναπτυγμένο οπουδήποτε στον κόσμο. Οπότε και εσείς και εγώ είμαστε κάπως πρωτοπόροι. Καμιά φορά στα οικονομικά υπάρχει αυτή η φράση της ε, ποινής που πληρώνει κάποιος να κάνει κάτι ε, πρώτος. Λοιπόν, ε, στόχος βεβαίω, η πρόεδρος διακόπτει τον κύριο Λέβη. Mm. Α, να καθίσω μάλιστα. Ε, θα έλεγα πως είναι μια εκτίμηση και όχι κασία για το κόστος ε, του οργανωμένου εγκλήματος ε, και βεβαίως να υπάρχει έτσι μια σωστή εκτίμηση κατάστασης για την Επιτροπή σας και τους υπόλοιπους. Είμαστε στην πρώτη φάση, υπάρχουν τρεις φάσεις ε, και στόχο έχει έτσι να δημιουργηθεί πρώτα απ' όλα ένα θεωρητικό πλαίσιο και αργότερα θα δούμε το δημοσιευμένο υλικό που υπάρχει στην Ευρώπη και αλλού και να αναπτύξουμε κάποιους τομείς που θεωρούμε εμείς ε, εφικτούς μαζί με τις επιφυλάξεις μας βεβαίως για την αξιοπιστία και τέλος θα καταλήξουμε στο που θεωρούμε ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα. Τώρα το αναλυτικό μας πλαίσιο θα είναι να διαχωρίσουμε τα δεδομένα σε ε, δεδομένα εγκλήματος ε, αγοράς θα έλεγα ή εγκλήματος με θύμα. Θα το δείτε αυτό μετά στα, στην Ιταλική έκθεση δηλαδή. Τέτοιο έγκλημα με θύματα είναι η κλοπή, η ανθρωποκτονία, διαρρήξεις, τέτοια πράγματα. Απάτη. Και βεβαίω υπάρχει και το οργανωμένο έγκλημα που απευθύνεται σε μια αγορά όπως ε, το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, ε, και η εμπορία ανθρώπων. Και βεβαίως ε, θα καταλήξουμε και στο άμεσο και έμεσο κόστος και το διαχωρίζουμε σε ιδιωτικό και μη κόστος. Ε, υπάρχει δηλαδή κάποιο κόστος ε, το οποίο διαχέεται σε ολόκληρη την κοινότητα, σε αυτούς που συνδέονται κατά κάποιον τρόπο με το έγκλημα. Δηλαδή αν συμβεί μια δολοφονία ή βιασμός σε μια κοινότητα, αλλά ε, όλοι όσοι γνώριζαν τα θύματα ε, εμπλέκονται πιο άμεσα από το κοινό γενικώ. Και βεβαίως ο έλεγχος προς τα πάνω και προς τα κάτω και το κόστος της αντίδρασης. Τι θέλω να πω λοιπόν, το κόστος ε, είναι μεγαλύτερο από το όφελος του εγκληματία. Βλέπουμε π.χ. σε εφημερίδες πως κάποιος δολοφονήθηκε ξέρω εγώ για ένα ευρώ. Είχε 10 ευρώ πάνω του. Και έτσι θεωρούμε πως είναι πιο τραγικό το έγκλημα. Ε, εδώ το κοιτάμε σε μεγαλύτερη κλίμακα. Αν δούμε όπως είπα τα, θύμα, τα εγκλήματα με θύμα π.χ. τιμωρία κάποιου ο οποίος δεν πληρώνει εκβιαστές, ε, προσωπικές απάτες, κλοπή μετάλλου που βλάπτει, πλήττει του σιδηρόδρομου σε ολόκληρη την Ευρώπη για να βγάλει κάποιος τώρα πενταροδεκάρες έτσι από τα καλώδια. Ναι. Ε, ηλεκτρονικές επιθέσεις ε, είναι αυτά στο παράρτημα της έκθεσής μου. Εκεί πέρα ε, το κόστος είναι μεγαλύτερο από το κέρδος του εγκληματία. Ε, Μπόριο ανθρώπων και βεβαίως απόρριψη τοξικών αποβλήτων. Όλα αυτά έχουν τεράστιο κόστος στην κοινωνία, πολύ μεγαλύτερο από το όφελος του ε, εγκληματία παρά το ότι όπως επεσήμανε ο από την Πολωνία ε, η κατάσχεση είναι ένα σημαντικό μέσο παρόλα αυτά ποτέ δεν θα μπορέσουμε να ανακτήσουμε τόσο πολλά ακόμα και να ξεχάσουμε το ότι οι εγκληματίες ξοδεύουν πάρα πολλά σε, σε γρήγορες γυναίκες και κουτσά άλογα όπως λέγεται ίσως ελαφρές γυναίκες και αργοκίνητα άλογα θα λέγαμε καλύτερα. Αλλά δεν θα μπορέσουμε ποτέ να καλύψουμε το κόστος ε, ε εγκλήματα όπως είπαμε αγορά αλλά και Εντάξει, Ίσως εκεί πέρα, ας πούμε, στο εμπόριο ναρκωτικών κάτι να γίνεται, αλλά όταν κάποιος αγοράζει πλαστά φάρμακα, δεν γνωρίζει ότι είναι πλαστά, έτσι. Ενώ ε, αν αγοράσει μια τσάντα από το δρόμο, και είναι ευθυνή, ξέρει πως δεν είναι γνήσια. Είναι, αν θέλετε, ένα συμβόλαιο για μια υπηρεσία. Οπότε, το κόστος μπορεί να είναι πρώτα απ' όλα απτό. Διαφθορά, βία, ή μία από το π.χ. η ανησυχία της κοινή γνώμης για την παράνομη μετανάστευση ή για νέους ε, που πέφτουν στα ναρκωτικά, το τζόγο ή την ε, πορνογραφία στο διαδίκτυο. Τα αποτελέσματα λοιπόν είναι μεγαλύτερα όταν δεν υπάρχει κάποιος στον οποίο μπορούν να απευθυνθούν τα θύματα για να διορθώσει την κατάσταση στην προσωπική και επαγγελματική τους ε, ζωή. Σε πολλά μέρη της Ένωσης ε, η κατάσταση βεβαίως διαφέρει. Δεν είναι παντού ίδια. Οπότε το να υπολογίσουμε το κόστος του οργανωμένου εγκλήματος ε, παρουσιάζει ένα πρόβλημα γιατί έχουμε πολύ μεγάλο μέρος της εγκληματικότητας ε, που εμπίπτει εντός του ορισμού της συνθήκης του ε, Παλέρμο. Δηλαδή τρία ή περισσότερα άτομα που συμφωνούν να κάνουν μια δραστηριότητα από κοινού για ε, μια περίοδο χρόνου. Οπότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το οργανωμένο έγκλημα ως εξής να δούμε δηλαδή τις μαφιόζικες οργανώσεις που πολλοί θεωρούν πως καταπιέζουν την κοινωνία, οι περισσότεροι δηλαδή πλήν των μαφιόζων ή το χαμηλότερου επίπεδου οργανωμένο έγκλημα, όπως ε, π.χ. δίκτυα ανθρώπων που μπορεί και να μην γνωρίζονται, αλλά συνεργάζονται με τρόπο εγκληματικό που οι περισσότεροι μπορεί να μην θεωρούν ε, οργανωμένο έγκλημα. Αλλά εμπίπτει εντό ε, του ορισμού της συνθήκης του Παλέρμου. Οπότε εάν αφήσουμε εκτός τις ε, απάτες που κάνουν μονομένοι απαταιώνες, που μπορεί να είναι από πολύ μικρές μέχρι πολλών εκατομμυρίων ευρώ, ε, η δεύτερη κατηγορία συμπεριλαμβάνει όλα τα εγκλήματα που διαπράττουν στην Ευρώπη για οικονομικό όφελος, συν το κόστος ε, που υφίσταται η κοινωνία για να ελέγχει την επικράτεια και βεβαίως το κόστος από τα παράνομα αγαθά. Ε, υπάρχει λοιπόν κάποια τυπολογία εδώ πέρα και συμπεριλαμβάνονται διάφορες ε, δραστηριότητες. Δεν θα μπω τώρα σε λεπτομέρειες, αλλά συμπεριλαμβάνει τα αναμενόμενα, συν ε, το περιβαλλοντικό έγκλημα, συν το έγκλημα εις βάρος της φύσης και το έχουμε αναλύσει με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή σε αυτούς τους τομείς. Και στην άλλη στήλη βλέπετε τα οργανωμένα εγκλήματα που προτείνω να αποκλείσουμε από τη μελέτη. Θα τα συζητήσουμε. Θα συζητήσουμε αυτά της αριστερής στήλης. Αλλά το ξέπλυμα χρημάτων, ηλεκτρονικό έγκλημα, διαφθορά, κλοπή ταυτότητα, και όλα αυτά είναι αυτό το οποίο η Europol, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ αποκαλούν αν θέλετε τις, ε, τα στηρίγματα του εγκλήματος γιατί αν συμπεριλάβουμε και το ξέπλυμα του χρήματος μετράμε δύο φορές τέτοια πράγματα. Μετράμε δύο φορές το κόστος δηλαδή. Ναι, ναι, γνωρίζω πόσο χρόνο πιέζει κυρία Πρόεδρε. Περνάω λοιπόν στο κόστος του εγκλήματος που σχετίζεται με τα ναρκωτικά. Θα είναι δύσκολο να γνωρίζουμε βεβαίως ποιο ποσοστό της ζημίας που προκαλούν τα ναρκωτικά πρέπει να αποδοθεί στο οργανωμένο έγκλημα. Ε, υπό μίαν έννοια όλος, όλο το κύκλωμα των ναρκωτικών αποτελεί αντικείμενο του οργανωμένου εγκλήματος. Οπότε όλη η ζημιά που προκύπτει είναι κομμάτι του κόστους του οργανωμένου εγκλήματος. Αλλά κάποιο από αυτό το κόστος, εν μέρη τουλάχιστον, είναι ζήτημα του πώς αντιμετωπίζουμε το έγκλημα και τους εγκληματίες και παρά το ότι τα ανώτερα επίπεδα της διανομής, εξαγωγής και χοντρικής πώλησης ε, ε, περιλαμβάνουν ε, περίπλοκες οργανώσεις, το χαμηλό επίπεδο είναι μεμονωμένοι πολιτές που εργάζονται για λογαριασμό τους, συχνά για να χρηματοδοτήσουν το δικό τους εθισμό είναι αν θέλετε έμποροι χρήστες ε, παρά άτομα τα οποία θα θεωρούσαμε ε, μαφιόζους. Δεν νομίζω καν πως εμπίπτουν στον ορισμό του Παλέρμου. Οπότε, να υπολογίσουμε το κόστος, κάτι οποίο θα κάνουμε το καλοκαίρι. Θα είναι κάπως ε, δύσκολο, αλλά βεβαίως θα δούμε τη χρήση κάποιων ε, παρανόμων ναρκωτικών. Θα δούμε βεβαίω την ε, ειδική κάναβη, τις αμφεταμίνες, ε, την κοκαίνη και την ηρωίνη. Και βεβαίως δεν είναι ακριβή τα στοιχεία, ούτε θα τα επινοήσουμε εμείς. Αυτό είναι το κόστος λοιπόν του εγκλήματος που σχετίζεται με τα ναρκωτικά. Ε, είναι μεγάλη η συζήτηση λοιπόν στην βιβλιογραφία για το ποιες ε, πτυχές ε, του κόστους πρέπει να εξετάζουμε. Π.χ. αν υπάρχουν τεκέδες μειώνεται το κόστος ή ε, εάν παρέχει το κράτος κάποιο, κάποιες δωρεάν ενέσεις και χώρους ίσως για ενέσεις, μειώνεται έτσι η μετάδοση του HIV. Εάν δούμε την απάτη, Βλέπουμε εδώ πέρα το κόστος ε, από πλευράς διαφθοράς ε, που μας αποσχολεί ιδιαίτερα, ε, καλά εμένα γιατί είμαι και στην Επιτροπή Διαφθοράς και συμβουλεύω και άλλου, αλλά δεν χρειάζεται τώρα να επανεφεύρουμε τον τροχό, αλλά θα εξετάσουμε και αυτά τα δεδομένα. αλλά το κόστος ε, βεβαίως αφορά και τους πολίτες και τους κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα εξετάσουμε επίσης ε, κεντρικά, την κεντρική, περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση, τον τομέα των κοινοφελή και άλλους τέτοιους φορείς, όπου πραγματικά η απώλεια εμπιστοσύνης στους κοινοφελείς φορείς ε, ως αποτέλεσμα της απάτης ε, επηρεάζει πάρα πολύ και το κατά πόσον ο κόσμος ε, κάνει δωρές. και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Η επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης επηρεάζονται. Υπάρχουν τεχνικά ζητήματα για, γιατί βεβαίως ε, το τι μπορεί να γίνει με θηγατρικές εταιρείες, ευρωπαϊκών εταιριών στο εξωτερικό και ή θηγατρικές αμερικανικών ε, στην Ευρώπη. Ξέρω πως είναι επίμαχο το ζήτημα, η Google και η Amazon ε, είναι στις ειδήσει τελευταία, παρά το ότι είναι κατά βάση αμερικανικές εταιρείες για λόγους ε, φορολογίας έχουν ε, έδρα κάπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λοιπόν περίπλοκο το ζήτημα αυτό, θα προσπαθήσουμε να το λύσουμε. Το κόστος ε, το οργανωτικό αντιμετώπισης της απάτης και βεβαίως το κόστος του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης, το κόστος της δίωξης δηλαδή, που μπορεί να προκύψει αν και όταν αποκτήσουμε Ευρωπαίο Εισαγγελέα. Όλα αυτά λοιπόν είναι πολύ σημαντικά. Κάποια δουλειά έχουμε κάνει στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά δεδομένα δεν είναι τόσο ανεπτυγμένα. Ας θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για την Επιτροπή σας και πραγματικά υπάρχουν τρεις διαστάσεις θα έλεγα βλάβης και κινδύνου. Υπάρχει το οικονομικό κόστος και ο αντίκτυπος που έχει στα θύματα και σε τρίτα μέρη που φοβούνται παραδείγματο χάρη ότι θα εξαπατήσουν, ότι θα τους κλαπεί η ταυτότητα. Υπάρχουν υποερωτήματα, δηλαδή μας ενδιαφέρει αν τα θύματα είναι μη πολίτες σημαντικά ζητήματα όπως ποια είναι τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των θυμάτων και ο αντίκτυπός τους. Ε, η Ευρώπη, όπως και κάθε άλλη χώρα ε, στον κόσμο, γυράσκει. Επίσης ε, είναι πιο βλαβερό για την κοινωνία το να είναι τα θύματα πιο ηλικιωμένοι, όπως εγώ ας πούμε, όταν δεν έχουν πλέον μπροστά τους όλη τους, ε, τη ζωή για να ανακτήσουν τα κλεμμένα ή όταν τα θύματα είναι πιο νέοι. Ένα ενδιαφέρον ερώτημα που έχουν παραμελήσει γενικά οι οικονομολόγοι, αλλά είναι σημαντικό. Κάνει διαφορά το να έχει κανείς ούτως ή άλλως ε, ελάχιστα και να πες θύμα απάτης ή αν έχει πολλά και χάσει περισσότερα λεφτά. Το επόμενο θέμα είναι το πώς παρουσιάζουν τα ΜΜΕ τους κινδύνους. Γνωρίζουμε όλοι, ακόμα και αν δεν ζείτε στο Ηνωμένο Βασίλειο, ότι γνωρίζουμε την διαστρέβλωση των συστημάτων του εγκλήματος και έτσι δημιουργείται μια νέα πραγματικότητα την οποία πρέπει να αντιμετωπίσετε εσείς ως πολιτικοί και εγώ ως πανεπιστημιακός. Μετά, άλλοι κίνδυνοι που προκύπτουν από αυτούς που διαπράττουν τα οικονομικά εγκλήματα. Υπάρχουν οργανωμένοι εγκληματίες που δεν έχουν ζήτημα ε, προσώπου που θα παρουσιάσουν στην κοινωνία και έχουν πρόσβαση σε προσωπικό το οποίο είναι πλέον πιο εκβιάσιμο ή ευεπίφορο σε διαφθορά, όπως είπε πρόσφατα, ειδικά σε καιρούς ε, ύφεσης, όπως είπε πρόσφατα ο Διευθυντής της ε, Europol. Δεν ξέρω κατά πόσον ισχύει αυτό το οποίο υπόθηκε πως ε, μόνο τα κονδύλια του εγκλήματος έχουν σώσει την Ευρώπη από την καταστροφή, αλλά τέλος πάντων μάλλον υπάρχει ένας αυξημένος κίνδυνος σε καιρούς ύφεσης. Οπότε Εμείς, ε, εμάς μας ζητήθηκε να σας δώσουμε μια εικόνα του κόστους του οργανωμένου εγκλήματος, αλλά ελπίζουμε να ε, αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς για το μέλλον, για τη ΛΥΜΠΕ και για άλλους, για την αξιολόγηση του εάν τα πράγματα χειροτερεύουν ή βελτιώνονται. Μπορεί να συμβεί και αυτό. Οπωσδήποτε πες ένα ζήτημα είναι το εάν τα πράγματα πάνε χειρότερα, αν γίνονται οι άνθρωποι πιο ευάλωτοι στη διαφθορά. Π.χ. στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Κάποιοι θα πούν πως ε, ήταν διατεθειμένοι να διαφθαρούν και πιο πριν αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά οπωσδήποτε άμα είναι να προσπαθούν να διατηρηθούν σε ένα επίπεδο διαβίωσης, ε, να είναι πιο ευάλωτοι στον πειρασμό. Και Εάν ο εγκληματίας ε, θεωρεί πως περισσότεροι θα μπορέσουν να δεχτούν ε, τις προτάσεις του, μπορεί να αυξηθεί η απάτη και το ξέβλημα χρήματος. Και το άλλο ζήτημα είναι πού ξοδεύουν τα λεφτά τους. Εάν δηλαδή μπαίνουν ξανά στις επιχειρήσεις ή ε, κάπου που μπορεί να κατασχεθεί όπως είπατε ή εάν πηγαίνει βεβαίως ε, ξοδεύεται σε γιορτές ε, δεν θα έλεγα πως αποταμιεύεται ας πούμε και υπάρχει κάποια προτεσταντική θα έλεγα ηθική. Άλλοι τομείς που μας απασχολούν είναι το κόστος της εμπορίας ανθρώπων που είπα πριν πως είναι σημαντικό. Βλάπτει βεβαίως ε, πάρα πολλούς. Βεβαίως η διαχωριστική γραμμή μεταξύ εμπορίας ανθρώπων και του όλου αυτού κυκλώματος ε, παράνομης μετανάστευσης είναι μπελεπτή. Βεβαίω ο κόσμος δεν θα πλήρωνε κιόλας για αυτή την υπόθεση αν θεωρούσε πως θα τον εκμεταλλευτούν. Και όχι μόνο αυτή, αλλά και στο μέλλον. Κινέζοι, Μολδαβοί και λοιποί δεν θα έδιναν μεγάλα ποσά για να μπουν στην Ευρώπη. Συχνά χρωστάνε, δεν χρωστάει η οικογένειά τους. Αλλά ε, δεν θα έδιναν τα ποσά αυτά εάν δεν ε, ανέμεναν πως θα βρουν κάποια δουλειά εδώ στην Ευρώπη για να ξεπληρώσουν τα δανεικά. Οπότε είναι σαφές πως... Εντάξει, είναι κόστος αυτό υπό μία ανένεια, αλλά το κόστος για τους Ευρωπαίους, ναι, δεν εργάζονται παράνομα, δεν πληρώνουν φόρους και τα λοιπά. Ναι, υπάρχει αυτή η πτυχή ε, του κόστους ε, εις βάρος ε, της Ευρώπης, αλλά ε, υποφελούνται οι οικογένειές τους στη χώρα τους. Δηλαδή αρκεί να δείτε μόνο τα εμβάσματα μέσω της Western Union και άλλων αναλόγων εταιριών για να καταλάβετε πόσο εξαρτώνται κάποιες χώρες εκτός της Ευρώπης από την παράνομη αυτή εργασία. Οπότε είναι περίπλοκο να υπολογίσουμε το κόστος της εμπορίας ανθρώπων. Δεν θα το θεωρήσουμε, όπως είπα, κάτι τελείως ε, καταπιστικό, γιατί παρά το ότι οι συνθήκες εργασίας είναι άσχημες, ε, μπορεί να είναι καλύτερες από αυτές που ισχύουν στη χώρα τους. Γι' αυτό πληρώνουν και για να έρθουν εδώ. Οπότε είναι εγκληματική η δραστηριότητα, σημαντική. Και θα προσπαθήσουμε να υπολογίσουμε το κόστος. Μετά, εγκλήματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ήδη έδωσα κάποια δεδομένα. Και αυτό κοστίζει. Παραχάραξη χαρτονομισμάτων. Και ανέφερα, όπως είπα, τα στηρίγματα αυτά του εγκλήματος, ηλεκτρονικού εγκλήματος, βία, διαφθορά κλπ. Θα τα δούμε διαφορετικά αυτά. Αυτά είναι κάποια παραδείγματα επίσης του πώς αναλύουμε τα εγκλήματα που έχουν θύματα. Δεν μιλάμε δηλαδή μόνο τις απώλειες αλλά και την ψυχική οδύνη κτλ. Και, και το πώς επηρεάζει την ζωή των θυμάτων. Οπότε, τα δεδομένα αυτά. Υπάρχουν κάποια δεδομένα για την, τον αντίκτυπο τον οικονομικό και τον ψυχικό του οργανωμένου εγκλήματος στα θύματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν υπάρχουν μέτρα για το πόσο ωφελούνται οι εγκληματίες και το ποιο ποσό θεωρητικά θα μπορούσε να κατασχεθεί. Αν θέλετε κάτι τέτοιο, αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Τέλος, το κόστος του οργανωμένου εγκλήματος δεν ε, Επαρκεί για σκοπούς δίωξης γιατί ο αντίκτυπος ε, των διαφόρων μέτρων ε, σε κάθε τύπο εγκληματικότητας ε, πρέπει να συνυπολογιστεί. Οπότε, όπως είπε ο κύριος Νιούτον Ντάν, αυτό το οποίο είπε για τη μετατροπή της Europol σε ένα ερευνητικό σώμα από ένα σώμα πληροφοριών και, να συνέβαινε κάτι τέτοιο, πρέπει να δούμε κατά πόσο θα, ε, μειωνόταν έτσι το, το έγκλημα. Η σύνδεση δηλαδή μεταξύ των επιχειρήσεων των διοκτικών αρχών και της μείωσης του εγκλήματος είναι κάτι το περίπλοκο. δεν το έχει δει ακόμα κανείς, ε, όχι μόνο η Επιτροπή σας, ε, κανένας ερευνητής στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για την υπομονή σας. Και αναμένω τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ κύριε καθηγητά. Θα δώσω το λόγο στον Νιώτον Τάνου. Ευχαριστώ, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας. Το θέμα είναι πότε θα τελειώσει. Έχετε τεράστια δουλειά μπροστά σας. Εμείς τερματίζουμε το φθινόπωρο. Θα έχετε κάτι μέχρι τότε για να συμπεριλάβουμε στην έκθεσή μας. Ή θέλετε ακόμα ένα-δυο χρόνια. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Αυτό το οποίο μας είπατε θα μας είναι ιδιαίτερα χρήσιμο. Και δεύτερον, για ένα δευτερεύον θέμα, μιλώντας για το μικρό έγκλημα, το οποίο δεν είναι οργανωμένο όπως το διεθνές, σε πάση περιπτώσει. Ίσως εδώ δεν κάνω κριτική σε αυτό που είπατε, απλά προσπαθώ να σας απαλλάξω από κάποια πράγματα. Το κομβικό ερώτημα που τίθεται εδώ, γιατί πρέπει να ενημερώσουμε το κοινό, είναι πόσο θα μας βοηθήσει να γλιτώσουμε χρήματα ένα ευρωπαϊκό FBI. Προσπαθούμε να δούμε ποιο είναι το κόστος λοιπόν του εγκλήματος και από ό,τι φαίνεται φτάνει σε εκατομμύρια εκατομμυρίων και έκπληνση χρημάτων και παραχαραγμένα προϊόντα. Είναι τεράστια τα ποσά, πραγματικά τεράστια και αν ας είμαστε γενναιόδοροι ας τους δώσουμε ένα προϋπολογισμό ενός δις κατέτος. Τεράστια ποσά. Και αν με το ένα δις μπορούν να μας γλιτώσουν το 1% των εκατομμυρίων εκατομμυρίων όπως είπα, τότε αξίζει τον κόπο. Ακόμα και αν δεν είναι απόλυτα αποτελεσματική. Νομίζω λοιπόν ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό να δούμε ότι η απόδοση της επένδυσης ε, μέσω της δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής αστυνομικής δύναμης θα ωφελήσει πάρα πολύ την Ευρώπη. Και γι' αυτό η πρότασή σας θα μας είναι χρήσιμη και πολύτιμη. Και εμείς σαν πολιτικοί πρέπει να πείσουμε το κοινό και τις λιθαργικές στη συγκεκριμένη περίπτωση ε, κυβερνήσεις για τη χρησιμότητα. Λοιπόν, επανέρχομαι στην πρώτη ερώτηση. Πότε θα μας δώσετε τα στοιχεία σας. Βάιλα. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Γνωριστήκαμε στο Βερολίνο σε, μια, σε ένα συνέδριο. Και χαίρομαι που ήρθατε και στις Βρυξέλλες. και έρχομαι κατευθείαν στα συμπεράσματά σας. Το ερώτημά μου είναι τι προσφέρει ένα ευρωπαϊκό FBI, ένας ευρωπαίος εισαγγελέα. Δεν υπαρκεί, νομίζω, θεωρώ εγώ έτσι, να καταπλημίσουμε μόνο σε εθνικό επίπεδο κάποια πράγματα. Για κάποιες πλευρές εγκληματικότητας ίσως, αλλά Ακριβώς ο τομέας οικονομικά εγκλήματα θεωρώ πως είναι απολύτως απαραίτητο να ξεκινήσουμε από εκεί να έχει μια ευρωπαϊκή αντιμετώπιση και ξεπλάγει από την προσέγγιση σας την απεσιόδοξη για το ότι δεν λέτε πως δεν ξέρετε τι θα προσφέρει. Το θέμα δεν είναι μόνο τα λεφτά. Που όπως ε, έλεγε η τα πάλι λεφτά θέλουνε. Εμένα με ενδιαφέρει ο αποτρεπτικός χαρακτήρας. Γιατί όποιος κάνει οικονομικά εγκλήματα εντός της Ευρώπης ε, και εκτός ε, μπορεί ε, να μην φοβάται τίποτα. Γιατί αν φεύγει κανείς από τη χώρα του που γνωρίζει την ομοθεσία και πάει σε μια άλλη όπου είναι πιο χαλαρά τα πράγματα, μπορούμε να, μπορεί να χρησιμοποιήσει τα λεφτά εκεί. Αλλά, εάν υπήρχε ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο που θα έχει και αρμοδιότητες συνεργασίας με τρίτες χώρες, ειδικά σε ζητήματα φορολογικών οάσεων και ξεπλήματος χρήματος, τότε θα έπαιζε και ένα σημαντικό αποτρεπτικό ρόλο. Τι άποψη έχετε γι' αυτό. Ευχαριστώ. Συνάδελφε Μάγερ, έχετε το λόγο. Θα συμφωνήσω με τους δύο προλαλήσαντες. Εγώ δεν θα μιλήσω τώρα για Ευρωπαϊκό FBI. Αλλά θα ήθελα να μας πείτε αυτό το οποίο ζήτησε και ο κύριος Νιούτον Ντάν. Π.χ. Europol έχει λίγα άτομα για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και πρέπει να ασχοληθεί με 27 χώρες. Και πρέπει να παίξει ένα ρόλο και εντός της Ένωσης αλλά και στον συντονισμό με άλλες χώρες. Γιατί μην ξεχνάμε και την απάτη του ΦΠΑ. η οποία ανέρχεται σε πολλά δισεκατομμύρια και σχετίζεται και με οργανωμένο ε, έγκλημα και μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλα ποσά και η Europol έχει 12 άτομα για αυτή την απάτη του ΦΠΑ. Οπότε θα έπρεπε νομίζω να υπάρχει στελέχωση έτσι ώστε τουλάχιστον να υπάρχει μεγαλύτερη προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλύτερος συντονισμός καταπολέμησης του εγκλήματος σε συνεργασία με τις εθνικές αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές. Ευχαριστώ. Ζόμπρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ήταν η παρουσίαση. Την παρακολούθησα με μεγάλο ενδιαφέρον. Έχω μία ερώτηση. Ίσως να το έχετε αναλύσει κι εσείς. Θεωρούμε προφανές ότι το έγκλημα παράγει κόστος. Κλοπές και άλλα εγκλήματα. Και αυτό είναι κάτι που μπορεί να αποστοτικοποιηθεί. Υπάρχει κι άλλο κόστος όμως, όπως απώλεια εμπιστοσύνης. Είναι μια άλλου είδου απώλεια. Σε μια κοινότητα, πραγματος χάρη, σε μια κοινωνία, οι πολίτες μπορεί να υποχρεωθούν να εγκαταστήσουν συναγερμούς και άλλα μέτρα προστασίας, συσκευές, και αυτό είναι κάτι που επηρεάζει και το επίπεδο της ζωής των πολιτών. Κυρίως αν αυτού του είδους τα εγκλήματα ε, είναι ευρέως διαδεδομένα. Άρα το έγκλημα προξενεί πολλές συνέπειες. Προξενεί και έμεσο κόστος, πέρα από το άμεσο. Αναλύσατε και το κόστος που προξενούν οι διάφορες συμμορίες και το πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα κλίμα που να αποτρέπει τους επιχειρηματίες από το να επενδύουν. Το βλέπουμε στην Πολωνία αυτό να συμβαίνει, στον τομέα των οικοδομών. έχει λάβει κονδύλια η Πολωνία για έργα υποδομής. Αλλά περίπου 200 εταιρείες στον τομέα των οικοδομών χρεοκόπησαν. Διότι δεν τους κατεβλήθησαν τα ποσά εγκαίρως. Αυτό είναι ένα γεγονός που έχει αποτρεπτικό αποτέλεσμα για τους επιχειρηματίες. Αυτό είναι κάτι που οδηγεί στην έλλειψη εμπιστοσύνης. Επηρεάζει επίσης την οικονομική ανάπτυξη και την οικονομική δραστηριότητα εν γέννη. Άρα έχουμε απώλεια εμπιστοσύνης που αυτό παράγει ένα κόστος. Υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης έναντι των δυνάμεων επιβολής της τάξεως και, του, και της δικαιοσύνης εν γέννη. Υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης εναντί των δικαστηρίων, των εισαγγελικών αρχών, που κανονικά είναι φορείς που κινούνται για την προστασία των πολιτών από το έγκλημα. Άρα οδηγεί σε αύξηση του κόστου από πλευρά πολιτών που θέλουν να προστατευθούν έναντι των φαινομένων. Εξετάσατε λοιπόν και το κόστος που συνεπάγεται η απώλεια της εμπιστοσύνης. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος ο κ. Γιακολίνο έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ακούσαμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, εκτός από το τελευταίο κομμάτι και ζητώ συγγνώμη, αλλά πράγματι εξετίμησα δεόντως τις θέσεις και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τα προβλήματα. Προβλήματα ευρωπαϊκού τύπου. Νομίζω ότι η ευρωπαϊκή πρόκληση ακριβώς θα μας οδηγήσει στο μέλλον να αξιολογήσουμε σωστά το κόστος των συστηματικών αυτών δικτύων που ε, παρανόμος ε, φύγουν με άμεσους και έμεσους τρόπους την πραγματική οικονομία. Αναφερθήκατε στα οργανωτικά πρότυπα και στο κόστος ε, αυτών των προτύπων. Δύο τίθενται εδώ τα ερωτήματα. Κατά πόσον επηρεάζει το κόστος ε, σε ποιο βαθμό, εν πάση περιπτώσει, η πραγματική οικονομία αμφισβητείται στην ουσία από την ύπαρξη αυτών των εγκληματικών δικτύων. Πολλές φορές η ανταγωνιστικότητα των τοπικών ιδιαιτέρως ε, οικονομιών ε, υπονομεύεται από την διείσδυση αυτών των παράνομων εγκληματικών συστημάτων. Ε, σε ποιο βαθμό μειώνεται η ανταγωνιστικότητα αυτών των περιοχών. Και δεύτερον, στα πλαίσια αυτής της προοπτικής πόσο θα βοηθήσει η γυτνίαση θα έλεγα των ευρωπαϊκών νομοθεσιών απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα και τη μαφία μέσω μιας διαδικασίας ενορμόνησης των νομοθεσιών και πόσο ε, θα βοηθήσει να μειωθεί το κόστος το οποίο προκαλεί η ύπαρξη των εγκληματικών αυτών δικτύων Σταδιακά βέβαια πρέπει να προχωρήσουμε γιατί προς στιγμή ε, δεν υπάρχει θα έλεγα μια συγκεκριμένη δυνατότητα. Τόμασιτς ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, καλωσορίζω και εγώ τον κύριο καθηγητή. Δεν θα ήταν φθηνότερο να διευκολύνουμε την καταπολέμηση της εγκληματικής δραστηριότητας προτείνοντας μηδενική ανοχή σε οποιονδήποτε έχει σχέση με το δημόσιο και έχει μια δημόσια θέση. Πολλά από τα εγκλήματα αυτά δεν θα μπορούσαν να συμβούν αν δεν υπήρχαν κάποιοι στο εσωτερικό του συστήματος. Για να καταπολεμήσουμε τη διαφορά απαιτείται μια πραγματικά αποτελεσματική δυνατότητα της ομάδας που θα την καταπολεμήσει. Ευχαριστώ κυρία Τόμασιτς. Ο κύριος Λεβί έχει το λόγο για να απαντήσει. Θα δούμε αν οι ερωτήσεις σας ήταν καλύτερες από τις απαντήσεις μου. Πολύ ενδιαφέρουσες οι ερωτήσεις σας και θα προσπαθήσω να απαντήσω με τη σειρά που τέθηκαν. Λοιπόν, τέλος Σεπτεμβρίου θα ολοκληρώσουμε ε, την εργασία, οπότε θα την έχετε. Δεν είναι πάρα πολύ ε, ο χρόνος για να ολοκληρώσει κανείς μια τόσο μεγάλη προσπάθεια, αλλά δεν είμαι μάγος, δεν μπορώ να εφεύρω ψευδή δεδομένα ή ψευδείς στόχους για να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις σας. Θα υπάρξουν κάποιες εκκρεμότητες σε σχέση με ορισμένα δεδομένα τα οποία δυστυχώς με μαγικό τρόπο δεν μπορούμε να εφεύρουμε μόνο και μόνο γιατί τα χρειαζόμαστε. Το θέμα της ε, δευτερεύουσας εγκληματικής δραστηριότητας ή της τοπικής εγκληματικής δραστηριότητας. Λοιπόν, αυτό άπτεται της γενικότερης προβληματικής σε σχέση με το επιτόπιο έγκλημα. Προφανώς ε, ένα σύστημα με, πυ, με πυραμίδες ε, μπορεί να λειτουργήσει τοπικά και ο κόσμος συνήθως χρησιμοποιεί για να πάρει μέρος σε αυτό το σχήμα πόνζι ε, τους φίλους του και τους γείτονές του για κάτι το οποίο πιστεύει ότι είναι ε, ωφέλιμο αλλά στο τέλος καταλήγει ε, σε μια απάτη ή αν γίνει μια δολοφονία η οποία φυσικά η δολοφονία επηρεάζει άμεσα αυτούς οι οποίοι κατοικούν σε μια συγκεκριμένη περιφέρεια. Υπάρχουν και κάποιες ερωτήσεις τις οποίες έθεσε η κυρία Βάιλερ σχετικά με το FBI και το πιθανό αποτρεπτικό ρόλο του ευρωπαϊκού σε εισαγωγικά FBI. Σίγουρα υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερη διαμεθοριακή δραστηριότητα των αστυνομικών δυνάμεων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εν την πλήρη αυτή έχει δημιουργήσει ένα πρόγραμμα για την χρήση ειδικών ανακριτικών ή ερευνητικών ε, αρμοδιοτήτων στον τομέα του οργανωμένου εγκλήματος και της ποινικοποίηση ορισμένων ενεργειών. Υπάρχει όμως ανάγκη για περισσότερες διαμεθοριακές ε, δραστηριότητες. Δεν ήμουν ιδιαίτερα σκεπτικιστής ως προς αυτό. Αυτό το οποίο προσπάθησα να πω στις τελευταίες μου παρατηρήσεις είναι ότι η μεθοδολογία για την σωστή κατανόηση της σχέσης ανάμεσα σε πόρους εκτός αστυνομικής δραστηριότητας και ε, ε, το τι μπορεί να κάνει η κοινωνία με λίγα λόγια εκτός από τις αστυνομικές ενέργειες για να μειώσει το οργανωμένο έγκλημα είναι κάτι που δεν έχουμε ακόμα εξερευνήσει δεόντως. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπάρχει ανάγκη για τη χρήση περισσότερων δυνατοτήτων και πόρων και πρέπει να γίνουν και περισσότερες ερευνητικές και ανακριτικές προτάσεις. Ίσως να είναι και 12 αυτοί στην Ευρωπόλ που ασχολούνται με τα θέματα αυτά, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί στα κράτη-μέλη. Πρέπει να βρούμε λοιπόν τρόπους έτσι ώστε να συνεργαστούν με καλύτερο τρόπο και στις χώρες ε, προέλευσης και στις χώρες, ε, αν θέλετε, κατάληξης της συγκεκριμένης έρευνας κάθε φορά. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι το οποίο με αφορά άμεσα. Εγώ θα συμφωνήσω πλήρως με αυτά που είπατε για τις απάτες στον τομέα του ΦΠΑ σαν παράδειγμα. Εγώ έκανα την διδακτορική μου εργασία πριν 40 χρόνια για την αντιμετώπιση των απατών μέσω των πτωχεύσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο τότε, αλλά είχα πει ότι πράγματι πρόκειται για μια εγκληματική διεθνή δραστηριότητα. Ήδη υπάρχουν νομοθετικές ρυθμίσεις ε, στον 16ο αιώνα ήταν έγκλημα το να εξαπατούν τους πιστωτές τους και το να διαφεύγουν στο εξωτερικό. Το φαινόμενο είναι γνωστό λοιπόν εδώ και πολλούς αιώνες, αλλά είναι κάτι που έχει πάρει πάρα πολύ μεγάλο μέγεθος και δεν υπάρχει σωστή δίωξη τέτοιου είδους συμπεριφορών. Όλοι βρισκόμαστε στην ίδια φάση και στο ίδιο επίπεδο, αλλά και θα συμφωνήσω εδώ ότι απαιτείται να υπάρξει κάποια, κάποια στοιχεία, να υπάρξουν κάποια στοιχεία αποτροπής έτσι ώστε οι πολίτες ούτε να νιώθουν ότι διώκονται αλλά δεν είναι και ε, θύματα αν θέλετε κάποιων μηχανισμών ε, α, ανάκτησης των χρημάτων τα οποία έχουν ε, αποκτήσει μέσω ποινικά κολάσιμων διαδικασιών στο παρελθόν. Το θέμα τώρα της εμπιστοσύνης εμείς θα προσπαθήσουμε ακριβώς να προτείνουμε μέτρα προς την κατεύθυνση της αύξησης του αισθήματος εμπιστοσύνης. Εδώ είναι δύσκολο να βάλει κανείς απόλυτα αριθμητικά στοιχεία. Έτσι κι αλλιώς εμένα τα απόλυτος αριθμητικά στατιστικά στοιχεία μου δημιουργούν κάποια δυστημία αυτοί οι οποίοι είναι σίγουροι για τα ποσοστά τους και βάζουν συγκεκριμένους αριθμούς σε ε, μη υλικέ αν θέλετε ε, ε, μορφές και δομές με κάνουν να είμαι επιφυλακτικός αλλά εδώ υπάρχουν και, τα, και οι δευτερεύουσες θα έλεγα ζημίες ακριβώς από την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών δηλαδή ζημίες για αυτούς που δεν ήταν ακριβώς ο πρώτος στόχος. Τώρα, για την μηδενική ανοχή σε αυτούς οι οποίοι εργάζονται για το δημόσιο. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό δεοντολογικό θέμα. Δεν νομίζω ότι η εγκληματολογία έχει να δώσει μία απάντηση ε, στο αν έχει σημασία αν έχει κανείς μηδενική ανοχή ή 0,5 ανοχή που λέει ο λόγος. Ε, μερικές φορές η επιδίωξη της απόλυτης ε, ακαιρεότητας οδηγεί δυστυχώς ε, σε μια ιεράρχηση πραγμάτων εκτός των σημαντικών. Και Νομίζω ότι η προσπάθεια που κάνουμε τώρα και εμείς και εσείς ε, μας βοηθούν για να δούμε πραγματικά ποια είναι τα σχετικά μεγέθη των εγκληματικών δραστηριοτήτων. Αν διώκουμε λοιπόν τους πάντες ακόμα και για πάρα πολλά ε, και πολύ μικρά ποσά, τότε δεν θα έχουμε και τους πόρους που απαιτούνται για να διώξουμε τα διασυνδεδεμένα εγκληματικά συστήματα όχι μόνο των ε, τεράστιων εγκληματικών ενεργειών, αλλά και αυτών οι οποίοι συμμετέχουν σε περίπλοκα δίκτυα. Αν χρησιμοποιήσει κανείς όλους τους πόρους που έχει στη διάθεσή του στα μικρά προβλήματα, τότε δεν θα έχει πόρους και δυναμικό για τα λύσει τα μεγάλα. Ε, δεν φαίνεται να σας ικανοποιούν αυτά που λέγω, αλλά εν πάση περιπτώσει αν έχεις δεδομένους πόρους θα πρέπει να αποφασίσεις πού θα τους στρέψεις. Είναι μια πολιτική πραγματικότητα αυτή, θλιβερή αλλά αληθής. Καμία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει όλες τις εκφάνσεις της εγκληματικότητας. Απαιτείται λοιπόν η ιεράρχηση και οι προτεραιότητες να καθοριστούν και αυτό το οποίο προσπαθώ να κάνω είναι να σας βοηθήσω να στραβείτε προς τα εκεί. Ακόμα και αν ε, υπακούει κανείς ε, σε ε, κανόνες και σε αρχές νομιμότητας όπως σε χώρες σαν την Ιταλία με το δίκαιό της, παρόλα αυτά θα πρέπει να αποφασίσει αν θα κυνηγήσει τα μεγάλα ψάρια όπως προσπαθεί η Ευρωπόλ ή τα μικρά που και αυτά ίσως θα πρέπει Φυσικά και είμαι θεωρητικά υπέρ της μηδενικής ανοχής, αλλά όταν ε, εκφράζει κανείς την μηδενική ανοχή ε, στον τομέα της, εγκλημα... της δίωξης της εγκληματικότητας, αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το εξετάσουμε προσεκτικά. Ευχαριστώ κύριε καθηγητά Λεβί. Θα πρέπει να θυμίσω ότι κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης των συντονιστών θα αξιολογήσουμε την δυνατότητα γνωρίζοντας ότι η τελική έκθεση δεν θα είχε φτάσει έγκαιρα για το σύνολο των εργασιών μας. Είχαμε κάνει όμως μια διαφορετική μορφή αξιολόγησης, είχαμε πει ότι υπάρχει ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε και να θέσουμε σε χρήση αν θέλετε την έκθεση αυτή και για την Επιτροπή μας. Περιμένουμε λοιπόν την τελική φάση της έρευνάς σας και θα τη στη διάθεση ε, του συνόλου της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ λοιπόν τον κύριο καθηγητή Λιβάη. Περιμένουμε τα τελικά αποτελέσματα. Ο Μπίλ. Yes. Ε, ε, ε, ναι. Σέβομαι τα όσα είπε η Πρόεδρος, ορθά ήταν. Μήπως μπορούμε να βρούμε κάποια δυνατότητα πριν την ψηφοφορία στην Ολομέλεια να ακούσουμε τον κύριο καθηγητή να μας κάνει μια μικρή παρουσίαση όσον αφορά τα πορίσματά του για να συζητήσουμε. Θα ήταν πολύτιμο αν τα καταφέρουμε. Θα ήταν πολύτιμο για όλους αν καταφέρουμε να γίνει κάτι τέτοιο. I am, uh, the final vote is... Η τελική ψηφοφορία είναι 9 Σεπτεμβρίου, λέει ο καθηγητής. 17. Στην Επιτροπή κοιτάξτε, θα προσπαθήσω να δω τι μπορώ να κάνω. Δεν έχω μαζί μου την ατζέντα μου και έχω και άλλες υποχρεώσεις αυτή την εβδομάδα στο Μεξικό όπου εκεί κάνω μια μελέτη τι μπορούν να κάνουν οι επιχειρήσεις για το οργανωμένο έγκλημα εκεί. Θα προσπαθήσω όμως να είμαι διαθέσιμος ή δυνατόν. Θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω κάποια στοιχεία και πριν από αυτή την ημερομηνία. Ευχαριστώ, καθηγητά Λίβα Πάμε στο τελευταίο πάνελ αυτής της συνεδριάσεως. Έχουμε τους εκπροσώπους της Ευρωπόλ που τους καλώ εδώ. Ο Μισελ Ρόσεμπαχ που είναι επιχειρήσης μονάδα των σοβαρών μορφών του οργανωμένου εγκλημάτων και τον κ. που είναι ειδικό για το οργανωμένο έγκλημα στην Ιταλία. Θα μας παρουσιάσουν χρησιμότατα στοιχεία προς προβληματισμό Όσον αφορά την πρόσφατα δημοσιευμένη έκθεση, όσον αφορά την εξολόγηση τη απειλή από πλευρά οργανωμένου εγκλήματο, του Ιταλικού οργανωμένου εγκλήματο, αναλύεται η εμβέλεια του οργανωμένου εγκλήματο, του διεθνού Ιταλικού εγκλήματο και τι απειλή δημιουργεί για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για τον υπόλοιπο κόσμο. Επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω, και αυτή είναι η προσωπική άποψη, ότι αυτή η έκθεση που θεωρώ προσωπικά ότι είναι εξαιρετικής σημασίας και εμβελίας και είναι ακρογωνίως λήθος των εργασιών μας και κάνει μια εποχιακή αναλύση του φαινομένου και ρίχνει το φως επί του προβλήματος που θεωρεί το περιφερειακό και εθνικό αρχικά και καταστρέφει το τελευταίο το πολιτιστικό εμπόδιο που υπήρχε επί σειρά ετών. Και το θερούσαν οι πολιτικοί και το χρησιμοποιούσαν διάφοροι πολιτικοί για να οχυρωθούν και να μην αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα και να μην εξετάσουν ε, εις βάθος το φαινόμενο αυτό του οργανωμένου εγκλήματος στην Ιταλία και των Ιταλικών εγκληματικών οργανώσεων. Όπως πάντα θα δώσουμε 20 λεπτά σε κάθε ε, φιλοξενούμενο, μετά θα διεξαχθεί συζήτηση με τη συμμετοχή των ε, συναδέλφων. Α, έκανα λάθος. 20 λεπτά συνολικά στη διάθεση των δύο μιλητών. 10 λεπτά για τον καθένα. Μετά θα υποβληθούν ερωτήσεις από τους συναδέλφους και ξανά θα δοθεί ο λόγος στους φιλοξενούμενους. Ο κύριος Μισελ Ρόσεμπαχ είναι ο πρώτος που θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ την Επιτροπή που κάλεσε την Ευρωπόλ σε αυτή την συνεδρίαση. Έχετε τους χαιρετισμούς του Διευθυντού Ρέπεν Ράιτο στην Επιτροπή. Λυπάτε που δεν μπόρεσε να παραστεί σήμερα στην Επιτροπή. Θα σας παρουσιάσουμε τα πορίσματα της Ευρωπόλ όσον αφορά την αξιολόγηση της απειλής που αντιπροσωπεύει το οργανωμένο έγκλημα το Ιταλικό. Ο κ. Ρέινρατ το συζήτησε το έγγραφο αυτό επανειλημμένα από την κυρία Αλφάνο και μου ανέθεσε ε, να την ευχαριστήσω για την υποστήριξή της ε, για το θέμα αυτό. Η Ευρωπόλ δεν ξεκίνησε αυτή την αξιολόγηση της απειλής πρόσφατα. Όχι μόνο αυτό, ε, ο Διευθυντής τον Μάιο πρόσφατα μαζί με τους επικεφαλής αστυνομίας της αστυνομίας ετοίμασαν ένα σημείο επαφής, είναι επιχειρησιακό πρόγραμμα που στοχεύει συγκεκριμένες ομάδες εγκληματιών και μορφές εγκλημάτων που εξετάζονται από την Ευρωπόλ. Έχει ξεκινήσει η δουλειά δηλαδή. Και ο κύριος Έλερο δίπλα μου διευθύνει την όλη επιχείρηση και την ομάδα και από τώρα και στο εξή θα παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυ το οργανωμένο έγκλημα ιταλικού τύπου στο μέλλον. Και ελπίζουμε ότι στο εγγύς μέλλον να μπορέσουμε να σας δώσουμε τα πρώτα πορίσματα. Πριν ξεκινήσουμε με την αξιολόγηση της απειλής, θα δώσω το λόγο, και πριν δώσω το λόγο στον συνάδελφο, να προβώ σύντομα σχόλια για το έργο της Επιτροπής. Η Ευρωπόλ θεωρεί ότι η Επιτροπή σας είναι σημαντικότατη διότι το οργανωμένο έγκλημα, η διαφθορά και το ξέπλυμα χρήματος είναι πολύ επιζήμια για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους πολίτες της και θα πρέπει να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για την εντόπιση του φαινομένου. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την αξιολόγηση του σοβαρού εγκλήματος ε, που ξεκίνησε η Ευρωπόλ πρόσφατα. Είναι λεπτομερέστατη προσέγγιση, λεπτομερέστατη αξιολόγηση όσον αφορά τι συνέπειες που έχει το οργανωμένο έγκλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τι είδαμε είδαμε ότι το οργανωμένο έγκλημα και ομάδες οργανωμένου εγκλήματος τύπου μαφίας παίζουν σημαντικό ρόλο στον τομέα του εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βάσει της σοβαρότητας του φαινομένου, το Συμβούλιο Εσωτερικών και Δικαιοσύνης έθεσε προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για την μετώπιση του προβλήματος για τα επόμενα χρόνια. Και αυτό δίνει μία πολιτική όθηση στην προσέγγιση και στις κοινέ δραστηριότητε που εφαρμόζουμε η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. Κάποιες ενδείξεις να δώσω όσον αφορά τα πορίσματά μας, όσον αφορά τα εξελόγηση του κινδύνου. Εντοπίσαμε και εκτιμήσαμε ότι υπάρχουν 3.600 εγκληματικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεγάλη αλλαγή βλέπουμε στη συμπεριφορά και τη σύσταση των ομάδων. Είναι παγκοσμίου εμβελία, δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι πιο ευέλικτε, προσαρμόζονται, εκμεταλλεύονται νομικά κενά και ανακατεύονται σε νέε αγορέ όπου βλέπουν ότι υπάρχουν ε, μεγάλα έσοδα, χαμηλό κίνδυνο είναι πολυτάλαντες, χρησιμοποιούν διάφορες μορφές εγκλημάτων, να χρειαστούν ειδικού τους πληρώνουν για συνεργαστούν, συνεργάζονται σε παγκόσμιο επίπεδο μεταξύ τους, αλλά έχουμε συνεργασία των εγκληματικών ομάδων. Αυτό ισχύει βέβαια και για τις Ιταλικές εγκληματικές ομάδες. Συνεργάζονται με εγκληματικέ μονάδες που κινούνται σε άλλους τομείς εγκληματικούς και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές του κόσμου. Είναι πολύ φευρετικές ομάδες, εκμεταλλεύονται ό,τι μπορούν για να διαπράξουν τα εγκλήματά τους. Ακριματαλεύω την οικονομική κρίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει σαφή σχέση μεταξύ της οικονομικής κρίσης ε, με το οργανωμένο έγκλημα. Και υπάρχει αντίκτυπος από πλευράς του οργανωμένου εγκλήματος όσον αφορά την οικονομική ανάκαμψη. Η διαφθορά ε, η απειλή, δημιουργία αρνητικού, κλίμα, αρνητικού κλίματος επηρεάζει αρνητικά το κλίμα. Και δεν τηρούνται οι κανόνες για τον τονικό ανταγωνισμό. Ε, μετά η παραχάραξη προϊόντων ε, είναι κάτι επιβλαβές για την εμπιστοσύνη των πολιτών και είναι επιβλαβής για τις ε, κανονικές εταιρείες. Και το εμπόριο λευκής αρκός ε, τροφοδοτεί τις ανάγκες για φθηνά εργατικά χέρια λόγω της οικονομικής κρίσης. Δεν κλέβει μόνο τους πολίτες οργανωμένο έγκλημα, αλλά και άμεσα από τους προπολογισμού των κρατών μελών. Παράδειγμα, απάτη στο ΦΠΑ. Πρόσφατα, η απάτη όσον αφορά το εμπόριο εκπομπών του άνθρακος οδήγησε σε απώλειες περίπου 5 δις ευρώ. Μετά φορολογικές ε, απώλειες 11 δις περίπου από απάτη στον τομέα των φορολογικών. Στην Ευρωπόλ βλέπουμε άμεσες απόλυσεις όσον αφορά τις πληθυντικές κάρτες. Το 2011 ήταν περίπου 1,3 δις ευρώ. Τόσο υπολογίστηκαν. Και γίνεται ένας φαύλος κύκλος. Δηλαδή η οικονομική ύφεση δημιουργεί ευκαιρίες και δυνατότητες για τις εγκληματικές οργανώσεις και το οργανωμένο έγκλημα από την άλλη με τι αστηριότητέ του εμποδίζει την οικονομική ανάπτυξη. Αυτό συζητήθηκε και πριν στην Επιτροπή αυτή και επηρεάζει και τους διαθέσιμους πόρους για την επιβολή του νόμου. Η απειλή του οργανωμένου έγκληματος δεν αναγνωρίζεται στο βαθμό που θα έπρεπε και γι' αυτό η Ευρωπόλ υποστηρίζει το σχέδιο εκθέσεως και τις συστάσεις της Επιτροπής. Είμαστε πεπισμένοι ότι θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταπόκρισης, απάντηση που θα δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο φαινόμενο και να μειωθούν τα αρνητικά αποτελέσματα την κοινωνία. Καλωσορίζει η Ευρωπόλ, ιδιαίτερα την έκκληση για νομοθετικέ προτάσει που θα έχει κοινού ορισμού όσον αφορά το οργανωμένο έγκλημα, θα συμπεριλαμβάνει και τα δίκημα τη συμμετοχή σε οργανώσει τύπου μαφία. Πιστεύουμε επίση ότι θα μπορούσαμε να αυξήσουμε την ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τι κατασχέσει σε περιουσία και σε μετρητό, διότι η μετακίνηση του ρευστού είναι το καλύτερο εργαλείο ε, για να ανακτηθούν τα παράνομα έσοδα. Όσον αφορά την ανάκτηση των στοιχείων ενεργητικού, πιστεύουμε ότι κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να έχει κεντρικό μητρό για τα πεζικούς λογαριασμούς και ενθαρρύνει τις διάφορες υπηρεσίες ανάκτησης των πόρων να ανταλλάσσουν ε, πληροφορίες με την Ευρωπόλ μέσω του ασφαλου συστηματο συστήματο ανταλλαγής πληροφοριών. Αυτές είναι μία-δύο προτάσει τη Ευρωπόλ και αν ενδιαφέρεστε με τα χαρά σα δώσουμε λεπτομερέστερε πληροφορίε γραπτώ. Πριν δώσω το λόγο στον συνάδελφό μου, τον David Ελέρο, που είναι ειδικό για το οργανωμένο έγκλημα ιταλικού τύπου, θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή σα για μία ακόμη φορά που μα μας καλέσατε συγγνώμη, και σα διαβεβαιώ ότι η Ευρωπόλ καταβάλει κάθε προσπάθεια μαζί με τα κράτη-μέλη για να καταπολεμήσει το οργανωμένο έγκλημα, κυρίως τις Ιταλικές εγκληματικές ομάδες. Ευχαριστώ πολύ και δίνω τώρα το λόγο στον κύριο Έλερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπω ότι υπάρχει και ρολόι στο τραπέζι, οπότε μπορώ να ελέγχω το χρόνο. Είμαι ο Ντέβιτ Έλερο, είμαι αξιωματούχος σε Ευρωπόλ, πριν από την εμπειρία μου στην Ευρωπόλ. Ήμουν, ε, ήμουν αξιωματικός της Ιταλική αστυνομία των Καραμπινιέ στην Ιταλία και θέλω να παρουσιάσω τα βασικά αποτελέσματα τη εξολογήσεως των απειλών που εξεπώνησε η Ευρωπόλ όσον αφορά το Ιταλικό οργανωμένο έγκλημα. Τι θα αναφέρω σήμερα. Πρώτα απ' όλα γιατί. Ποιο είναι το ιστορικό για τον αφορά το έγγραφο. Λοιπόν, πώς δημιουργήθηκε ε, αυτό το έγγραφο, ποια είναι τα ευρήματα αυτής της προσπάθειας και τι μπορεί να κάνει η Ευρωπόλ για να προχωρήσουμε από εδώ και πέρα. Ήδη από το 2012 στα πλαίσια της προηγούμενης αξιολόγησης καταλήξαμε στο ότι υπήρχε μία θα έλεγα ποινική δραστηριότητα, ποινικά κολάσιμη εννοώ, η οποία προέρχεται από το νότο της Ιταλίας υπήρχαν πάρα πολλά εγκλήματα τα οποία είχαν διαπραχθεί και γενικά είχαμε διαπιστώσει ότι υπήρχε και μία θα έλεγα περιορισμένη αναφορά στις δραστηριότητες αυτών των εγκληματικών ομάδων εκτός τουλάχιστον Ιταλίας. Αυτό μας οδήγησε στην ανάγκη να αξιολογήσουμε σωστά την απάτη, την κατάσταση και να προσπαθήσουμε να την κατανοήσουμε καλύτερα. Από πλευράς των δυνάμεων καταστολής πάντα εννοώ. Όπως είπε και ο κύριος Ράσενμπακ, δημοσιεύθηκε η αξιολόγηση του 2013. 6.200 εγκληματικές ομάδες εντοπίστηκαν ότι λειτουργούν στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Ράσενμπακ αναφέρθηκε σε αυτά. Το βασικό θέμα το οποίο θα έλεγα ε, είναι ότι υπάρχουν κάποιες ήμι παράνομες δραστηριότητες ή δραστηριότητες διείσδυσης μη ομάδων σε νόμιμες ε, τουλάχιστον κατόνομα δραστηριότητες. Η μεθοδολογία μας τώρα, ε, στείλαμε ερωτηματολόγια στα διάφορα κράτη-μέλη και στις τρίτες χώρες με τις οποίες έχουμε συμφωνίες συνεργασίας. Οι ερωτήσεις είχαν σχέση με τον τρόπο λειτουργίας αυτών των εγκληματικών ομάδων και δυστυχώς ένα από τα πρώτα πράγματα που ήρθε στην επιφάνεια ήταν η έλλειψη ενημέρωσης για τις ομάδες αυτές εκτός των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούνται. Λόγω ακριβώς λοιπόν αυτής της έλλειψης ε, αναγκαστήκαμε να χρησιμοποιήσουμε τις διαθέσιμες πηγές και επίσης και τα εντάλματα τα οποία είχαν ήδη εκτελεστεί εις βάρος ε, Ιταλών εγκληματιών. Υπήρξε ένα δημόσιο κείμενο το οποίο μπορεί να διαβάσει οποιοδήποτε στην ιστοσελίδα μας και υπάρχουν επίσης και κάποιες πιο απόρριτες μορφές του εγγράφου που έχουν αποσταλεί στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Η αξιολόγηση των απειλών τώρα ξεκινάμε με μία σύντομη παρουσίαση της φύσης λειτουργίας και φύσης αυτών των ομάδων. Δεν ήταν αυτός ο βασικός μας στόχος βέβαια. Ο βασικός μας στόχος ήταν να δούμε πώς επηρεάζουν οι ομάδες αυτές όταν λειτουργούν εκτός της χώρας τους, η διεθνής τους διάσταση δηλαδή. Προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε τις βασικές Ιταλικές ομάδες, Κοζανόστρα, Ντράγκετα, Καμόρα, αλλά και ε, οργανωμένες ομάδες της απουλίας ε, όπως η Διστήτα. Καλύπτουμε επίσης και κάποιες άλλες ζώνες άσκησης της εγκληματικής δραστηριότητας Αυτού του είδους η εγκληματική δραστηριότητα δεν είναι κάτι το οποίο στοχεύει θα έλεγα έναν συγκεκριμένο κλάδο θα έλεγα παρανομίας αλλά ε, πηγαίνει παντού και προσπαθεί όπου μπορεί να έχει κέρδη να δραστηριοποιείται φυσικά ναρκωτικά το βασικό το μεγαλύτερο ναρκωτικά ε, πλήσιμο βρώμικου χρήματος ε, φυσικά διαφθορά που διευκολύνει τα πάντα ε, παραχαραγμένα προϊόντα, τοξικά απόβλητα και σωματεμπορία. Αλλά δεν σταματούν εδώ, είναι, είναι τεράστιος ο, ο αριθμός των δραστηριοτήτων της παρανομίας αυτής. Αυτό το οποίο έχει επίσης πολύ μεγάλη σημασία είναι οι τάσεις. Στις διαφάνειες βλέπετε εδώ ε, το τι είπε ένας από τους εισαγγελείς που πήρε μέρος στις συναντήσεις μας τον προηγούμενο Δεκέμβριο. Ε, τα οργανωμένα εγκλήματα, οι οργανωμένες ομάδες αν θέλετε αντιμετωπίζουν τα αντίθετα προβλήματα από τις ε, ε, νόμιμες αν θέλετε οργανώσεις οικονομικών συμφερόντων. Έχουν πρόβλημα ρευστότητας οι, οι, επιχειρηματικές ομάδες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ έχουν το αντίθετο πρόβλημα οι εγκληματικές ομάδες οι οποίες αναζητούν τρόπους να ξεπλύνουν τα, τα κέρδη που έχουν, τα τεράστια ποσά και να τα νομιμοποιήσουν και αυτή είναι η βασική απειλή που έχουμε από πλευρά τους. Υπάρχουν και κάποιες ε, τάσεις επενδύσεων στον λεγόμενο πράσινο ε, τομέα της ε, βιομηχανικής δραστηριότητας και ταυτόχρονα το διαδίκτυο παρέχει νέες δυνατότητες στο οργανωμένο έγκλημα. Ε, ποια είναι λοιπόν τα συμπεράσματα της συγκεκριμένης έκθεσης. Ε, το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης σε σχέση με τη δραστηριότητα αυτών των εγκληματικών ομάδων. Υπάρχει ένα άνισο επίπεδο συνειδητοποίησης του βάρους αυτών των ομάδων. Στην Ιταλία φυσικά λόγω της παράδοσής μας και λόγω των δύσκολων στιγμών της ιστορίας μας έχουμε μια σε βάθος γνώση για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι ομάδες αυτές όταν όμως κανείς βγαίνει από την Ιταλία υπάρχει πολύ χαμηλό επίπεδο γνώσης και ενημέρωσης για τις ομάδες αυτές. Αυτές οι ίδιες οι ομάδες οι εγκληματικές βέβαια λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο ε, στο εσωτερικό της Ιταλίας και ε, εκτός αυτής. Ε, στις περιοχές από τις οποίες προέρχονται έχουν πάντα τον πλήρη έλεγχο του εδάφους τους ακόμα και σε επίπεδο στρατιωτικής ισχύω θα έλεγα. Όταν όμως κινούνται εκτός Ιταλίας έχουν ένα πολύ χαμηλό προφίλ, είναι πάρα πολύ διακριτικές και εδώ τίθεται το θέμα αν θέλετε της έλλειψης ενημέρωσης. Επειδή έχουν χαμηλό προφίλ και επειδή κάνουν εισοδισμό στην πραγματική οικονομία περνούν απαρατήρητες. Και αυτό είναι το βασικό σημείο απειλής που αντιπροσωπεύουν σήμερα. Αυτό μας οδηγεί λοιπόν στις συστάσεις της έκθεσης της Ευρωπολής Υπάρχουν αρκετές συστάσεις, ανείχνευση αν θέλετε, των και ταυτοποίησης αυτών των εγκληματιών που λειτουργούν εκτός Ιταλίας, φυσικά η, η διαμήραση και κατανομή πληροφοριών, φαίνεται να υπάρχει αν θέλετε κάποια προσπάθεια α, καταπολέμησης νομοθετικής της μαφίας στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν αναφέρομαι μόνο στην Ιταλική αντίληψη για τη λέξη μαφία εδώ, για το Ιταλικό οργανωμένο έγκλημα, αλλά αυτό καλύπτει όλες τις μαφιόζικου τύπου εγκληματικές ομάδες, γιατί οι ομάδες αυτές όταν βρίσκουν θα έλεγα παραθυράκια στην νομοθετική ρύθμιση στις διάφορες χώρες μέλη τα εκμεταλλεύονται αντιμετώπιση των κερδών αυτών των εγκληματικών δραστηριοτήτων. Ε, πολλές φορές μπορούμε να τους συλλάβουμε, να τους βάλουμε στη φυλακή, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο ανήκει στην καθημερινότητά τους, δεν τις επηρεάζει ιδιαίτερα. Όταν όμως τα περιουσιακά του στοιχεία τους κατάσχονται, τότε αυτό είναι κάτι που τους θίγει πραγματικά. Και ταυτόχρονα θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την υπάρχουσα εμπειρία, να την εκμεταλλευτούμε. Όπως είπα υπάρχουν χώρες, αναφέρθηκα στην Ιταλία, αλλά δεν είναι η μόνη στην Ιταλία η οποία έχει με πολύ αποτελεσματικό τρόπο αντιμετωπίσει τέτοιου είδους οργανωμένες εγκληματικές ομάδες. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπους έτσι ώστε να βασιστούμε στις θετικές εμπειρίες, τα θετικά παραδείγματα για να κάνουμε προτάσεις και λύσεις και στις υπόλοιπες χώρες που ζητούν τη στήριξή μας. Λοιπόν, ποια ήταν η απάντηση της Ευρωπόλ σε όλα αυτά. Την ίδια στιγμή που καταλήξαμε στον καθορισμό της απειλής, ταυτόχρονα εμείς δημιουργήσαμε μια εξειδικευμένη δομή για να αντιμετωπίσουμε το Ιταλικό οργανωμένο έγκλημα. Δημιουργήθηκε ένα focal point στις 3 Μαΐου με την πλήρη ενθουσιώδη στήριξη των Ιταλικών αρχών και των αστυνομικών αρχών και των δικαστικών ταυτόχρονα και άλλων 7 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η συμμετοχή κάποιων τρίτων χωρών επίσης, το Eurojust επίσης συμμετέχει σε αυτό το focal point γιατί απαιτείται και η καταστολή αλλά και η δικαστική εξουσία και η Interpol φυσικά είναι μια πάρα πολύ σημαντική οργάνωση η οποία μας επιτρέπει να έχουμε επαφές με χώρες με τις οποίες δεν έχουμε διμερείς συμφωνίες. Ε, ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι αυτού του Focal Point. Είναι μια πλατφόρμα για να βοηθά τις ερευνητικές διαδικασίες. Μέχρι τώρα η Αεροπόλ έχει στηρίξει τις Ιταλικές έρευνες, αλλά ποτέ ε, ασχολούμενη με τη συγκεκριμένη εγκληματική ομάδα, αλλά με το αντικείμενο της δραστηριότητάς της. Τώρα λοιπόν προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε και τα θέματα των, πολιτικών, των εγκληματικών αυτών οργανώσεων. Συνεργαζόμαστε φυσικά και με τις δυνάμεις καταστολής άλλων χωρών. Έτσι και αλλιώς η αξιολόγηση του κινδύνου την οποία έχουμε κάνει δείχνει ε, το, τη στρατηγική συνεισφορά μπορούμε να έχουμε στην καταπολέμηση αυτών των δραστηριοτήτων και επίσης ε, και σωστή ενημέρωση για τους μη Ιταλούς ε, διοκτικούς μηχανισμούς και από τότε που ξεκινήσαμε τη λειτουργία αυτού του focal point έχουμε βοηθήσει και μια πολύ μεγάλη ε, προσπάθεια επιχείρηση καταπολέμησης μιας οργανωμένης ομάδας η οποία όμως εξελίσσεται σε αυτή τη φάση και ως εκ τούτου δεν μπορώ να σας πω τίποτα περισσότερο. Λοιπόν έχω ένα λεπτό στη διάθεσή μου Περιέργως έμεινα στα χρονικά όρια τα οποία μου δώσατε. Είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ. Ξεκινάει η συζήτηση. Δίνω το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Γιακολίνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ακούσαμε τον κύριο Ελέρο και σίγουρα συμφωνούμε. Αυτά που ακούσαμε με αυτά που κάναμε το 15 μήνο των δραστηριοτήτων μας. Υπάρχει ταύτιση βούληση. θέλουμε συνεργασία. Εκτιμήσαμε και την απλή γλώσσα με την οποία αναφερθήκατε. Είναι πολιτικό πρόγραμμα αυτό η αντιμετώπιση της μαφίας. Και μέσω τη σύσταση αυτή τη επιτροπή το αναγνώρισε το Κοινοβούλιο ότι χρειάζεται αντιμετώπιση, είμαστε στο δρόμο. Δεν υπάρχει διαβεστησία στα κράτη-μέλη. Ε, υπάρχει διαφορετική ευαισθησία από ό,τι στην Ιταλία. Και δεν υπάρχει το ίδιο επίπεδο επίγνωσης παντού. Κάτι που διαπιστώσατε στις δραστηριότητές σας στα διάφορα κράτη-μέλη. Πρόκληση είναι ευρωπαϊκή, άρα χρειάζεται προσέγγιση νομοθετικών προσεγγίσεων, καλύτερη χρήση της κατάσχεσης, κυρίως προληπτικά. Και να μην υπάρχουν αμφιβολίες στα κράτη-μέλη. Για να αντιταχθούμε στη μαφία πρέπει να αφαιρούμε τους πόρους, τα αγαθά τους, τα παράνομα έσοδα των δραστηριοτήτων τους. Να επιστραφούν στην νόμιμη οικονομία. Ε, χαιρόμαστε διότι στις 3 Μαΐου προβλέφθηκε η κίνηση της δραστηριότητα να γίνει επιμερισμός των πληροφοριών μεταξύ 7 κρατών μελών με Ευρωπόλ, Eurojust, Interpol για να καταλήξουμε στην ελευθερία και την ασφάλεια που θέλουμε. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις μου. Είναι και ενθάρρυνση να προχωρήσετε. Θα δείτε και την έκθεσή μας ότι όσον αφορά τα δικήματα που περιγράψατε, περιβαλλοντικού χαρακτήρα, ότι ευθυγραμμιζόμεθα. Θέλω να ακολουθήσουμε τον ίδιο δρόμο. Θέλουμε να κινηθούμε προς την κατεύθυνση της ασφαλείας και της ελευθερίας των πολιτών. Ευχαριστώ κύριε Γιακολίνο. Ο κύριος Κίρκοπ έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις θα ήθελα να κάνω και τους αναφέρατε. Και τις δύο, οπότε δεν είναι τίποτα το καινούριο. Το πρώτο ερώτημα αφορά τη σχέση μεταξύ Europol και τοπικών αστυνομιών. Θεωρώ πως ε, όπου έχουν ε, αναλυφθεί πρωτοβουλίες υπάρχουν κάποιες δυσκολίες και τομέας αυτός σε σχέση με την τοπική αστυνομία είναι πως υπάρχουν περιπτώσεις όπου η αστυνομία η ίδια πρέπει να εξεταστεί πολύ προσεκτικά πριν περάσουμε σε, σε ουσιαστικές συζητήσεις. Αναρωτιέμαι τι σχέση βρήκατε στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Και το θέμα είναι πως αναφέρατε το ζήτημα του οργανωμένου εγκλήματος και τις δραστηριότητες στα όρια της νομιμότητας. Επειδή υπάρχουν πολλές νόμιμες επιχειρήσεις όπου οι ίδιες οι επιχειρήσεις δεν γνωρίζουν ε, ποιος τους ελέγχει. Που, που, το ότι δηλαδή τα λεφτά προέρχονται από εγκληματίες. Σε ποιο βαθμό λοιπόν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορους μηχανισμούς για να υπάρξει κάποια σύνδεση αν θέλετε για να αποφύγουν αυτό το πρόβλημα οι νόμιμοι επιχειρηματίες. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Α. Ναι. Και τώρα κύριος Μπίλ Νιούτον έχει το λόγο both of you for very interesting. Ευχαριστώ και τους δύο για τις ε, παρουσιάσεις αυτές ενδιαφέρουσες και πολύτιμες. Ε, τέσσερις-πέντε Ιταλικές οργανώσεις που μας περιγράψατε σε μεγάλη λεπτομέρεια είναι οι μεγαλύτερες συμμορίες από τις 3.600 που αναφέρατε σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι η Ιταλία έτσι η καλύτερη και μεγαλύτερη ή υπάρχουν και άλλες ε, που θα πρέπει να γνωρίζουμε. Μία ερώτηση είναι αυτή. Έτσι για, να καταλάβω τι γίνεται γενικώ. Και δεύτερον, η πολύ καλή αυτή συμβουλή πως πρέπει να καταλήξουμε στον ορισμό του εγκλήματος του να νίκει κανείς σε μαφιόζικη οργάνωση. Μα, κοιτάξτε, εμείς δεν είμαστε Ιταλοί. Ε, για, για, εμάς η λέξη μαφία σημαίνει κάτι συγκεκριμένο. Ενώ εσείς λέτε πως πρέπει να είναι ένας γενικός όρος. Μήπως να ευθύσουμε μια διαφορετική λέξη αντί για τη λέξη μαφία, γιατί η υπόλοιπη Ευρώπη δεν καταλαβαίνει τι εννοείται. Ε, πρέπει να βρεθεί μια άλλη λέξη, δηλαδή να πούμε οργανωμένη συμμορία μαφιόζικου τύπου, κάτι τέτοιο. Γιατί υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης. Και πράγματι έχετε δίκιο, δεν αναφέρονται αυτά τα ζητήματα στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και έχουμε πάρα πολλή δουλειά που να κάνουμε και σας ευχαριστώ και για την ε, παρουσίασή σας. Κύριε Σολμαίρ Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για αυτά τα οποία μας είπατε, πολύ ενδιαφέροντα επανερχόμαστε βλέπω συνεχώς στην Ιταλία. Κοιτάξτε, εμείς δεν συνορεύουμε με την Ιταλία, αλλά έχουμε οργανωμένο έγκλημα. Ειδικά στις μεθοριακές περιοχές ε, με την Τσεχία. Και την ανάλυση του πώς, παραδείγματος χάρη, ε, βιετναμέζικες ε, συμμορίες ε, έχουν εισχωρήσει και επηρεάζουν και την Τσεχία και την ε, χώρα μας. Οπότε το ζήτημα, το ερώτημα που ήθελα να θέσω είναι τι γίνεται με τη συνεργασία με κάποιες ασιατικές ε, κυβερνήσεις για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και συμμοριών που παραδείγματος χάρη στέλνουν τα λεφτά από τις εγκληματικέ δραστηριότητες στην Ευρώπη και τονώνουν ε, την ε, τοπική οικονομία ε, με χρήματα τα οποία βεβαίως έχουν βγει με βαριά, από βαριά εγκλήματα στην Ευρώπη. Και είναι δύσκολο λοιπόν να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος μετά. Το ερώτημα λοιπόν είναι χρειάζεται και συνεργασία στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής ε, και όχι μόνο της ε, αστυνομικής πτυχής για να υπάρχει και μια ανταπόκριση από πλευράς ε, π.χ. της βιετναμέζικης κυβέρνησης γιατί μας το έχει πει και η κυβέρνησή μας ότι δεν υπάρχει διάθεση συνεργασίας από πλευράς ε, του Βιετνάμ παραδείγματος χάρη. Ευχαριστώ Μπορσελίνο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Ευρωπόλ. Είναι σημαντικότατο το έργο της και άκρος ενδιαφέρον. Η αξιολόγηση της απειλής. Διερωτώ με, γιατί η αξιολόγηση της απειλής μόνο το 2013 ή το 2011 από ό,τι κατάλαβα ξεκίνησε ήδη. Διότι στο αξιολόγηση της απειλής έπρεπε να έχει προληπτική, προληπτικό χαρακτήρα. Αυτή η μελέτη, αυτή η αξιολόγηση, αν είχε γίνει πριν σήμερα στην Ευρώπη θα υπήρχε διαφορετική επίγνωση. Ακριβώς αναφερόσα στην έλλειψη επίγνωσης που στην Ιταλία την βρήκατε. Το ίδιο θα συνέβαινε και στην Ιταλία. Η παρουσία της μαφίας θεωρεί σαν κάτι που αφορούσε τον Νότο και η υπόλοιπη Ιταλία, η Βόρεια Ιταλία κυρίως υποτιμούσε το πρόβλημα και το θεωρούσε ότι είναι πρόβλημα μόνο αυτών των περιοχών των Νότιων. Μετά με ή χωρίς επίγνωση είδε ότι είχε μπει και είχε εγκατασταθεί και στην οικονομία και στις άλλες περιοχές η μαφία, κυρίως η Ντράγκετα και νομίζω ότι είναι πιο διαδεδομένη ε, και στην υπόλοιπη Ευρώπη λόγω της ιδιαιτερότητας των δραστηριοτήτων της. Ρωτώ, αν είχε γίνει πριν κατά την άποψή σας αυτή η εξολόγηση, σήμερα θα υπήρχε διαφορετική ευαισθητοποίηση στην Ευρώπη, θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε διαφορετικά το πρόβλημα ή θα ήταν σαν να ξεκινήσουμε από το έτος 0, όπως και τώρα. Ε, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ευχαριστώ κυρία Μπορσελίνο. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στους καλυμμένους. Ευχαριστώ τους ε, αξιωματούχους της Ευρωπόλ. Ε, η δουλειά τους ήταν πάρα πολύ σημαντική για την Επιτροπή μας. Ευχαριστώ και τον Διευθυντή Wen Wright που πάντα ήταν διαθέσιμος στα αιτήματά μας ε, και πριν τα αιτήματα που κάναμε για την έκθεση του οργανωμένου έγκλημα του 2011 και για μένα, πώς να το πω, είναι λίγο αργά που γίνεται αυτό του είδους η δουλειά. Διότι αυτό που έλεγε η κυρία Μπορσελίνο ήταν σωστό. Εμείς στην Ιταλία πραγματικά είχαμε παρατηρήσει μακρόν μία υποτίμηση, μία προσέγγιση επιφανειακή από πλευράς των πολιτικών και ίσως να εκπροσωπούσε και κάποιο συμφέρον, να μην βάλουν χέρι ε, να μην επηρεάσουμε μια νομοθεσία και να μην βρούμε μια απάντηση τεχνική και πολιτική. Άρα ξαναζούμε αυτό που ήδη ζήσαμε στην Ιταλία κατά το παρελθόν. Όταν όλο ήταν χαρακτηριστικό προνόμιο ίσως των περιοχών του Νότου και δεν λάμβαναν υπόψη ότι αυτό που συνέβαινε στο Νότο ήταν απλώς πρώτο τμήμα που αυτό που θα οδηγούσε σε επενδύσεις και κατάσταση στη Βόρεια Ιταλία. Είναι κάτι που βλέπουμε συμβαίνει ε, εδώ και πολλούς μήνες. Υπήρχε λοιπόν υποτίμηση ότι συνέβαινε μόνο σε μερικές περιοχές και αποσπάτω η προσοχή. Λοιπόν, συνέβη το ίδιο επιμακρών, δηλαδή ο όρος μαφία δεν εντοπίζει την Κόζα Νόστα, πούμε. Υπάρχουν διάφορες μορφ, ομάδες εγκληματικές, υποδιαιρούνται εδαφικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι οργανώσεις που έχουν έδρα την πουλια κινούνται μόνο στην πουλια. Έχουν ε, και άλλα συμφέροντα σε άλλες περιοχές της Ιταλίας. Το ίδιο ισχύει για την Κόζα για την Καμόρα, και για την Τράγκετα. Η Τράγκετα είναι η οργάνωση ισχυρότερη στον κόσμο πιθανότατα. Μη λησμονούμε όταν στην προηγούμενη συνεδρίαση ο εισαγγελέας Κατέρη λεπτομερώς μας παρουσίασε τις δυνατότητες που έχει η Ντραγκέτα να ξεπερνά τα όρια τα ευρωπαϊκά, να ευρεώνεται και να, δημιουργεί σχέσεις με το εμπόριο ναρκωτικών, ε, τους εμπόρους ναρκωτικών της Κολομβίας και με τους Μεξικανούς. Και τις προάλλες συνελήφθη ε, μία από τις πιο σημαντικές ε, ε, σημαντικά μέλη στην Κολομβία της οργάνωσης αυτής. Λοιπόν, αυτή μετακίνησε τρίτες χώρες, επέτρεψε σε διάφορες ομάδες. Όχι μόνο κάτι που αφορά την Ιταλία. Μιλάμε για ένα ευρύ φάσμα ομάδων. Με τον όρο μαφία συμπεριλάβουμε τις αστηριότητε των οργανώσεων των εγκληματικών στην Αφρική. Στην Ιγυρία, συζητήσαμε την Ιγυρία, ρωσικές μαφίες, ε, κινέζικες μαφίες, γιαπωνέζικες. Η Τισιόκα, ε, Μάλλον τον Ιούνιο του 2011 ο ίδιος ο πρόεδρος Ομπάμα αναφέρθηκε στο πρόβλημα. Αναφέρθηκαν τέσσερις τουλάχιστον εγκληματικές οργανώσεις που απειλούν τους Αμερικανούς πολίτες. Προτεραιότητα έχει η Ιαπωνέζικη μαφία και η Καμόρα. Όταν πήγαμε στη Ουάσιγκτον τον Απρίλιο, τέλος Απριλίου, αρχές Μαΐου, αναφερθήκαμε στην ανάγκη της μη υποτίμησης από πλευρά των οχών της ΥΠΑ των δραστηριοτήτων της Δραγκέτα. Δεν είναι κάτι που αφορά μόνο την Ιταλία. Εδώ συγκεντρωθήκαμε στην πραγματικότητα, στην κατάσταση της Ιταλίας για να μην υπάρξει μια υποτίμηση του φαινομένου. Αλλά ας πούμε η δραστηριότητα της δραγκέτας στη Γερμανία είναι κάτι υποδειγματικό. Παράδειγμα, έκαναν οργανωμένη, μελετημένη επίθεση κατά του κοινωνικού και οικονομικού ιστού της Γερμανίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει υποστεί εισβολή η Γερμανία από τη μαφία, αλλά υπήρξε μια υποτίμηση που επέτρεψε απεικιοκράτηση ομάδων από την Καλαβρία μελών της Δαγκέτα να ριζώσουν στην επικά της Γερμανίας και να συνεχίσουν να κάνουν τη δουλειά τους και να ε, επεκτείνονται. Σας ευχαριστώ για τη δουλειά που κάνατε. Για μένα είναι θεμελιώδου σημασία η δουλειά που κάνατε και το λέω. Ελπίζω να ληφθεί μια υποχρέωση, να πραγματική από πλευρά των κρατών μελών, να δραστηριοποιηθούν, να επενδύσουν ε, υπέρ της Ευρωπόλ, διότι η Ευρωπόλ είναι μια δομή που μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση. Αυτό εξαρτάται από τις πραγματικές προθέσεις όμως των κρατών μελών. Είδαμε πώς η Ευρωπόλ έθεσε στη διάθεσή μας μια σημαντικότητα δραστηριότητα. Ε, την έθεσε στη διάθεση αυτού του κοινοβουλίου, αυτού του φορέα. Αν γίνει η ίδια ανταλλαγή με τα κράτη-μέλη, να υπάρξει σωστή ροή πληροφοριών. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό κυρίως μέσω των εργασιών της Ευρωπόλ. Και όλα αυτά πρέπει να βγουν, οι προσπάθειες να βγουν από το πεδίο των πολιτικών δηλώσεων και να ελοπιθούν. Θα δώσω το λόγο στους δύο εκπροσώπους της Ευρωπόλ για να απαντήσουν στις ερωτήσεις και στα σχόλια των συναδέλφων. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Προς τον κύριο Γιακολίνο. Ναι, οπωσδήποτε. Μιλάει Ιταλικά, ναι. Εάν ήταν να ζωγραφίσουμε κάποια εικόνα, νομίζω πως ήταν, είναι σαφές αυτό το οποίο είπατε. Δηλαδή, οπωσδήποτε κατά την άποψή μου, έχουμε ένα ε, μαφιόζικο έγκλημα, το οποίο είναι διαφορετικό από το οργανωμένο έγκλημα. Και αυτό, ε, αυτή είναι η δυσκολία με την επικοινωνία εκτός Ιταλίας, γιατί όταν είναι να πείσουμε διοκτικές ε, δυνάμεις ε, να επενδύσουν ε, σε μια διοκτική επιχείρηση πρέπει να υπάρχει κάποιο αδίκημα έτσι και κάποιο αδίκημα στην Ιταλία η ύπαρξη μαφιόζικης οργάνωσης είναι ήδη αξιόπινη αλλά δεν υπάρχει αυτό σε άλλες χώρες πρέπει να έχει διαπρακτεί κάποιο άλλο έγκλημα Καταλάβατε. Οπότε αυτό αποτελεί βάση μέχρι να αναγνωριστεί λοιπόν ε, το ότι η μαφιόζικη οργάνωση είναι διαφορετική από το οργανωμένο έγκλημα θα έχουμε πρόβλημα. Και μετά ακολουθεί η υπόλοιπη αποτελεσματική στρατηγική και τα υπόλοιπα βεβαίω τα οποία λέτε τα δέχτηκε η Europol. Τώρα θα ήθελα να περάσω τον κύριο Κέρκοπ. Ελπίζω να προφέρω σωστά το όνομά σας. Πρώτο θέμα το οποίο είπατε, πώς ερχόμαστε σε επαφή με αστυνομικέ ε, δυνάμεις. Κοιτάξτε, υπάρχουν εθνικές μονάδες η Europol σε κάθε χώρα. Οπότε, όταν ε, έχουμε κάτι το οποίο αξίζει να ερευνηθεί, ερχόμαστε σε επαφή με την εθνική ομάδα, η οποία κανονικά ε, σε γενικές γραμμές, είναι σε επίπεδο υπουργικό, ε, λέει ποια είναι η αρμόδια αστυνομική υπηρεσία. Και μετά αντιστρόφως ε, ρέουν και οι άλλες πληροφορίες. Δηλαδή η τοπική αστυνομική δύναμη έρχεται σε επαφή με την εθνική ομάδα, την εθνική μονάδα και αυτή μετά με την Europol. Οπότε για μας είναι εύκολο να παρακολουθήσουμε τη ροή των πληροφοριών. Βεβαίω κανένα σύστημα δεν είναι τέλειο, αλλά νομίζω πως μέχρι στιγμής είχαμε θετικά αποτελέσματα. Το δεύτερο ερώτημα είναι πολύ ενδιαφέρον. Μιλάμε για νόμιμες επιχειρήσεις. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Και πράγματι μπορεί εκατοντάδες άνθρωποι να εργάζονται σε εστιατόρια, σε πιτσερίες που δεν ξέρουν ότι ε, ε, ξεπλένουν χρήμα. Αυτό σχετίζεται με μία σύσταση που κάνουμε στην έκθεση, γιατί πάρα πολύ συχνά ε, κάποιες ομάδες δεν γνωρίζουν το τι γίνεται, δεν μοιράζονται πληροφορίες, οπότε ναι βεβαίως, εάν κάποιος δεν πάει σε μια άλλη χώρα και τους πει προσέξτε λίγο γιατί αυτή η πιτσερία, αυτή η εταιρεία ή το οτιδήποτε σχετίζεται με ομάδα οργανωμένου εγκλήματος, στην άλλη χώρα δεν ξέρει κανείς τίποτα. Γιατί ο άλλος ανοίγει μια επιχείρηση. Έτσι, όταν βγαίνουν εκτός Ιταλίας δε, φοράνε τη γαβατούλα τους και εμφανίζονται σαν επιχειρηματίες. Οπότε, ε, σε χώρε θεωρούν πω ο κίνδυνο αυτό είναι πολύ χαμηλό κάτι το οποίο σχετίζεται με αυτό το οποίο είπε η κυρία Μπορσελίνα. Αυτή ήταν η κατάσταση στην Ιταλία πριν 20 χρόνια. Αυτό το οποίο πρέπει να αντιληφθούμε και πάντα λέω είναι πω σήμερα αυτοί οι άνθρωποι έρχονται με λεφτά, με πόρου σήμερα, έτσι, τη σήμερα ημέρα. Και μπαίνουν, ανοίγουν την πόρτα με τα λεφτά. Αυτή τη στιγμή εγκατασταθούν και εμφανίζονται ως επιχειρηματίες, μετά από λίγο καιρό θα έρθουν και οι εγκληματίες. Αλλά σε αυτή τη φάση αν έχουν ήδη εγκατασταθεί είναι πολύ δύσκολο μετά να τους εφορτωθείς, αν όχι αδύνατον. Αν μου επιτρέπετε δηλαδή να μιλήσω και ως καραμπινιέρος, το ίδιο είχε συμβεί στην Ιταλία πριν 20 χρόνια. Ε, εγώ είμαι από τη Βενετία έτσι γνώμη έλεγαν τότε μα δεν γίνονται τότε αυτά τα πράγματα στη Βενετία γιατί εμείς είμαστε αλλιώς όχι όχι αυτό είναι κοινή παρεξήγηση Κοίταξε έγινε στην Ιταλία έτσι αυτό, μιλάμε την ίδια γλώσσα. Ε, σκεφτείτε να πάνε σε τελείως διαφορετικές χώρες και πλαίσιο της Ευρώπης, όπου ο κόσμος δεν έχει ιδέα ε, τι είναι αυτό το πράγμα, έχει δει μόνο κάτι ταινίε στην τηλεόραση. Και αυτό σχετίζεται με αυτό το οποίο έλεγα για εκπαίδευση και πείρα. Πρέπει να εκπαιδεύσουμε, αυτός είναι ο δικό μας ο ρόλος, τις ευρωπαϊκές αστυνομίες για να αναγνωρίσουν τα σημάδια, για να σταματάνε αυτούς του ανθρώπους πριν εγκατασταθούν. Γιατί ε, βέβαια άμα, είναι, άμα περάσουν τα χρόνια μετά είναι πολύ αργά. Ελπίζω να απάντησα στο ερώτημά σας. Θα δώσω τώρα το λόγο στον ε, κύριο Αφενταχ. Ράσονταχ. Αν μου επιτρέπετε. Να σχολιάσω τα θέματα των συμμοριών αυτών και του μεγέθους τους. Ποια είναι τα μεγαλύτερα σχήματα, οι μεγαλύτερες συμμορίες. Καταρχάς, η απειλή την οποία θέτουν ε, αυτές οι οργανωμένες ομάδες εγκληματικές δεν καθορίζεται από από το μέγεθός της μόνο, από τον αριθμό των μελών της. Έχουν υπάρξει ίσως στο παρελθόν και μεγαλύτερες αριθμητικά ομάδες ανάμεσα στις 3.600 τις οποίες προανέφερα. Αυτό το οποίο είδαμε όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι έχει αλλάξει η εικόνα του οργανωμένου εγκλήματος και είναι πάρα πολύ δύσκολο να ορίσει κανείς ποιος είναι μέλος και ποιος ο οποίος ε, συνεργάζεται, συνδέεται με κάποιο τρόπο και είναι δύσκολο να βάλει κανείς την ε, ε, γραμμή τη διαχωριστική. Ποιος είναι μέλος και ποιος εργάζεται, συνεργάζεται, λειτουργεί σαν υπεργολάβος ή περνάει παράνομα κόσμο στα σύνορα σαν παράδειγμα. Όλα αυτά αλλάζουν συνεχώς. τη μία χρονιά έχουν κάποιους συνεργάτες, την επόμενη έχουν άλλους συνεργάτες σε μια ε, νέα αρχιτεκτονική ε, της λειτουργίας της ομάδας τους. Είναι δύσκολο να τα ορίσει κανείς όλα αυτά. Πάντως μπορούμε να πούμε είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται επιχειρηματικά αυτές οι ομάδες ε, είναι δύσκολο να τις κανείς γιατί προσαρμόζονται στις ανάγκες και στις δυνατότητες που παρουσιάζουν οι αγορές. Σχετικά με τα ονόματα η κυρία Αλφάνο αναφέρθηκε σε αυτό. Έχει σημασία να γνωρίζουμε γιατί μιλάμε, έχει σημασία να συνειδητοποιούμε το τι ακριβώς συμβαίνει και ήδη ε, συζητήθηκε από τους συναδέλφους. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι αυτές οι νέες μορφές οργανωμένου εγκλήματος δεν επηρεάζουν άμεσα τον πολίτη, όχι πάντα τουλάχιστον. Αν δείτε ας πούμε το θέμα της παραχάραξης ή τις μεγάλες απάτες για το ΦΠΑ, θα δείτε ότι επηρεάζονται έμεσα οι κυβερνήσεις. Οι κυβερνήσεις βέβαια, ε, οι πολίτες, συγγνώμη, οι κυβερνήσεις δεν έχουν τα μέσα για να αντιμετωπίζουν όλα αυτά. Γι' αυτό λοιπόν έχει σημασία να συνειδητοποιήσουμε όλοι με σωστό τρόπο τι είδος οργανώσεις είναι αυτές, τι φύσης οργανώσεις είναι αυτές. Και ανέφερε και ο κύριος Έλερο ότι η δύναμη ε, οφείλεται στις τεράστιες οικονομικές δυνατότητες που έχουν αυτές οι ομάδες, στους τεράστιους πόρους που έχουν αυτές οι ομάδες. Και εδώ αυτό που θα μπορούσε να παίξει ρόλο είναι η κατάσχεση των περιουσιακών του στοιχείων. Τώρα και εδώ έρχομαι στο πολύ δύσκολο ερώτημα που έθεσε η κυρία Χολμάια σχετικά με τις ασιατικές χώρες. Κοιτάξτε το νομικό μας πλαίσιο δεν μας επιτρέπει άμεσα να συνεργαστούμε με επιμέρους χώρες με τις οποίες δεν έχουμε συνάψει διμερείς συμφωνίες. Αυτό είναι κρίμα πολλές φορές γιατί εμείς φτάνουμε στα σύνορά μας και μετά πρέπει να δούμε άλλους τρόπους για να συνεργαστούμε με χώρες είτε μέσω των κρατών μελών είτε μέσω της Ιντερπόλ. Είναι δύσκολο όμως να έχουμε τις άμεσες επαφές οι οποίες απαιτούνται για να είναι κανείς ε, αποτελεσματικός. Ε, έχουμε συλλέξει ελάχιστες εμπειρίες. Ε, uh, uh, είναι λίγες εν πάση περιπτώσει οι περιπτώσεις στις οποίες μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις. Υπήρξαν κάποιες επιτυχεί, αν θέλετε ε, προσπάθειες και απόπειρε, αλλά όχι για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε γενικά συμπεράσματα. Ξέχασα μία ερώτηση. Ο κύριος Έλερο. Αυτό θα έπρεπε να είχε γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά όμως εγώ πήγα στην ε, Europol το 2007. Ε, δούλευα στην Νάπολη όταν πήγα εκεί και ήμουν υπεύθυνος για τα θέματα σώματεμπορίας. Το πρώτο θέμα που πήρε η Europol για την Ιταλία μας εστάλει το 2011. Ήταν η πρώτη περίπτωση που η Ευρωπόλ για πρώτη φορά ασχολήθηκε με το Ιταλικό οργανωμένο έγκλημα. Μα ζητήθηκε από την Ιταλία, πόσο μάλλον από άλλες χώρες βέβαια. Βέβαια όταν η Αεροπόλ, ξέρετε για τον κύκλο της ανταλλαγής πληροφοριών, όταν εμείς καθορίζουμε ορισμένες πληροφορίες ή μάλλον προτεραιότητες βασιζόμαστε στις πληροφορίες. Όταν το 90% των πληροφοριών αφορούν ας πούμε τα παραποιημένα προϊόντα, εμείς ε, προφανώς ασχολούμαστε με αυτό. Όταν πήγα στην Ευρωπόλ δεν υπήρχε ενημέρωση για τη δραστηριότητα των εγκληματικών ομάδων στην Ιταλία. Καθόλου. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Έλλειψη συνειδητοποίηση του προβλήματος εκτός Ιταλίας. Ίσως. Πολλές φορές ε, κάποιες αστυνομικές δυνάμεις δεν σκέφτονται να ενημερώνουν την Αεροπόλ. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Όταν αρχίσαμε να παίρνουμε στοιχεία και αυτό συμπίπτει και με την έναρξη της λειτουργίας της δικής σας Επιτροπής, τότε αρχίσαμε να έχουμε περισσότερα όπλα αν θέλετε στη διάθεσή μας και μπορούμε να πούμε ότι κοιτάξτε υπάρχει θέμα, υπάρχει πρόβλημα, ασχολείται και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να συνεργαζόμαστε με τις χώρες προέλευσης των στοιχείων. Η Γερμανία υποστηρίζει ιδιαίτερα τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία γιατί έχουν και αυτοί δύσκολες εμπειρίες σε σχέση με το Ιταλικό οργανωμένο έγκλημα. Έπρεπε να είχαμε ξεκινήσει πριν από πάρα πολλά χρόνια βέβαια και τότε θα ήταν αλλιώς η κατάσταση, αλλά δυστυχώς αυτά ε, διαφεύγουν του δικού μας ελέγχου. Ελπίζω την επόμενη φορά που θα έρθω να μιλήσω στο Κοινοβούλιο να μπορέσω να σας πω κάποιες επιχειρηματικές επιτυχίες, ε, επιχειρησιακές συγγνώμη επιτυχίες ε, που είχαμε, αλλά προς το παρόν είναι λίγο νωρίς και δεν μπορεί κανείς να διεκδικήσει κάποια νίκη. Ευχαριστώ. Ε, θέλατε να πείτε κάτι παρακαλώ. Δεν θα μιλήσω 25 λεπτά, αλλά έχουμε 25 λεπτά. Και καλό είναι που είναι εδώ πέρα οι mm. κύριοι για το σχόλιο περί εκπαίδευσης και των τοπικών αστυνομιών. Πραγματικά συμφωνώ στην εκλογική μου περιφέρεια. Πριν από κάνα δύο χρόνια ήμουν με ε, με μία από τις αστυνομίες της περιοχής μου. Και εκεί πέρα υπήρχε ένα κομμάτι χαρτί που έλεγε τηλέφωνα ξένων αστυνομιών. Και λέω ενδιαφέρον. Και ξένες αστυνομίες τι εννοούσανε δίπλα του Μάντσεστερ και του Νότιγχαμ στην αστυνομία. Οπότε ε, λες εκεί πέρα, δηλαδή απελπίζεσαι. Ε, πράγματι χρειάζεται εκπαίδευση. Ε, οι επαγγελματίες, οι, οι ειδικοί. Τι ξέρω πώς τους λέτε τους ανθρώπους αυτούς που δουλεύουν μεταξύ των, των συμμοριών, οι σύνδεσμοι αν θέλετε. Αυτή, αυτή είναι πραγματικά ισχυρή. Δεύτερο ερώτημα. Αυτά τα τεράστια κονδύλια που έχουν αυτές οι οργανώσεις. Πού είναι, κάτω σε κάποιες τράπεζες θα είναι. Ξέρουμε σε ποιες τράπεζες. Σε ευρωπαϊκές τράπεζες. Μήπως ε, σώζουν τους ισολογισμούς των Ευρωπαϊκών Τραπεζών. Και τέλος, σωστά είπατε, πρέπει ε, η ενημέρωση να προέλθει από πάνω προς τα κάτω. Και έτσι, που, έτσι όπως λειτουργεί η Ευρώπη πρέπει 28 αρχηγοί κυβερνήσεων να πούν τώρα αυτό είναι προτεραιότητα και πρέπει να κάνουμε κάτι σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το πώς θα γίνει αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά πρέπει να κινητοποιηθεί η κοινή γνώμη Γι' αυτό ο ρόλος αυτής της Επιτροπής είναι πάρα πολύ σημαντικός, γιατί δεν ξέρω αν μας δείχνουν ακόμα στο ίντερνετ, αλλά ελπίζω να μας ακούει κανείς. Εάν η κοινή γνώμη πει, μα δεν κάνετε τίποτα, είναι γελία η κατάσταση, κάνετε κάτι, τότε ε, μπορούμε να θέσουμε το θέμα στους 28 πρωθυπουργού και να γίνει κάτι. Ε, αυτή είναι η πραγματική πρόκληση. Πώς οι ηγέτες ε, θα κινητοποιηθούν για να αναλάβουν δράση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ξεκινήσω με την τελευταία σας ερώτηση. Πράγματι, μα γι' αυτό είμαστε εδώ. Γι' αυτό και δημοσιεύσαμε ε, μέρος της έκθεσης. Ε, αλλά αυτό δεν αφορά μόνο την, την κοινή γνώμη και για τις ε, αστυνομικές δυνάμεις που λέτε που θεωρούν το Μάντσεστερ εξωτερικό. Ε, το, Κοιτάξτε, μπορεί όταν ψάχνουν για καμιά δουλειά στο site της Europol να δουν και την έκθεση και να τη διαβάσουν και μου έχει συμβεί τρεις φορές. Παίρνουν τηλέφωνα από κάτι μικρές πόλεις και μου λένε κοιτάξτε πράγματα. Άνοιξε και εδώ πέρα ένα Ιταλικό εστιατόριο, είναι πολύ ευγενικοί όλοι, δεν έχουν κανένα πελάτη αλλά το μαγαζί είναι ανοιχτό. εκεί πέρα χτυπάει ένα καμπανάκι και έτσι ξεκινάνε τα πράγματα. Ξεκινάει μια έρευνα, καταλήγουν σε συλλήψεις και τα γράφουν οι εφημερίδες και τα διαβάζει ο κόσμος στι εφημερίδες και λέει κοίτα να δει που είχαμε τη μαφία και δεν το ξέραμε. Αυτά είναι γνωστά. Έχω ξάδερφο Άγγλο, ήταν ε, ε, σε ένα... Ήταν κάπου στην Αγγλία και καταδικασμένος μαφιόζος εκεί πέρα ε, Ιταλικό εστιατόριο και δεν θα, δεν θα το φανταζόταν ποτέ. Οπότε πραγματικά πρέπει να τεθεί το, το ζήτημα στο, στο κορυφαίο επίπεδο, στο πολιτικό. άλλο θέμα η εκπαίδευση. Τα, τα σημάδια δηλαδή που πρέπει να αναγνωρίζει κανείς, τα σημάδια της διείσδυσης. Γιατί αν δεν ξέρει κανείς ακριβώς τι πρέπει να κοιτάξει, μπορεί να, κοιτά, να, να ζητά κάτι τελείως διαφορετικό. Εάν, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν αυτές οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με μετρητά, εστιατόρια, πιτσαρίες, ε, δουλεύουν με πολύ μετρητό ένα βασικό σημάδι, ένα εύκολο πράγμα μπορώ να σου πω. Κοιτάξτε, εάν είναι μονίμως άδειο το μαγαζί και είναι ανοιχτό, λειτουργεί 10 χρόνια, από κάπου βγάζουν λεφτά αυτοί οι άνθρωποι. Για τα περιουσιακά στοιχεία. Πάρα πολλά. Κοιτάξτε, αν δείτε την Καλαβρία πολύ φτωχή περιοχή, αλλά οι εγκληματίε είναι από του πιο πλούσιου στον κόσμο. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι δημιουργούν φτώχεια στην περιοχή. Πού πάνε λοιπόν τα λεφτά. αυτό είναι το ερώτημα. Κάποια επενδύονται σε ακίνητα, γιατί τα ακίνητα θεωρούνται ακόμα ως ένα καλός τρόπος να μπουν τα λεφτά στην νόμιμη οικονομία. Βεβαίω, κομμάτι των χρημάτων ε, επανισάγεται στο τραπεζικό σύστημα. Αλλά τότε είναι ανοιχνεύσιμο, έτσι. Οπότε το σημαντικότερο κομμάτι μετά εμφανίζεται, δηλαδή οι μεσίτες, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι επισήμως θα έλεγα δεν είναι μαφιόζοι, αλλά δημιουργούν τον πλούτο τους, αυτό το οποίο λέμε την κρίζα ζώνη στην Ιταλία. που είναι για μένα ένα από τα πιο επικίνδυνα κομμάτια του οργανωμένου εγκλήματος. Γιατί? Γιατί όταν μπουν στην νόμιμη οικονομία, να αγοράσουν μετοχές, ξέρω εγώ, μιας εταιρείας. Αυτό που τους ενδιαφέρει δεν είναι η ίδια η εταιρεία, είναι το κύκλωμα σχέσεων στην νόμιμη οικονομία που έχει η εταιρεία αυτή. Αν μπουν π.χ. σε ένα franchise ή σε μια εταιρεία πληροφορικής. Ε, έρχονται σε επαφή με δικηγόρους, με συμβολεογράφους, με επενδυτές. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που δημιουργούν τον πλούτο των μαφιόζικων οργανώσεων. Κοιτάξτε, καμιά φορά μπορεί να είναι ενσωματωμένοι στη μαφία. Δηλαδή, Μπορεί κάποιοι ιδιαίτερο έξυπνοι να κάνουν μόνο σε αυτά τα πράγματα. Σε κάποιε περιπτώσει απλά παρέχουν υπηρεσίε. Και υπηρεσίε γενικώ στο οργανωμένο έγκλημα, όχι μόνο στο ιταλικό οργανωμένο έγκλημα. Να δούμε παραδείγματος χάρη γραφεία που στέλνουν λεφτά στο εξωτερικό. Υπάρχουν κάποια που είναι στην ιδιοκτησία τέτοιων ανθρώπων και Εάν ε, κάποιοι θέλουν να ξεπλύνουν χρήμα, πάνε τα λεφτά σε αυτούς και το ξεπλένουν αυτοί και κρατάνε ένα ποστό του χρήματος και παρέχουν μια υπηρεσία. Και αυτό δεν σχετίζεται οπωσδήποτε με ιταλικό ή ρωσικό έγκλημα. Είναι έγκλημα από μόνο του. Μάλιστα, το ΙΟΚΤΑ 2013 αναφέρει το ξέβλημα χρήματος ως ε, βασικό βασική προτεραιότητα και κάποιες ομάδες ειδικεύονται σε αυτό. Οι υποθέσεις τώρα στη Europol που έχουμε δει μέχρι στιγμής. Πράγματι υπάρχουν κάποιες τράπεζες που εμπλέκονται αλλά οι υποθέσεις ε, εκκρεμούν. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Ποιο είναι το βασικό δίδαγμα εδώ πέρα όμως για εμάς. Είναι πως ε, όσο καλή και αν είναι η νομοθεσία οι άνθρωποι αυτοί είναι επαγγελματίες πάντα θα βρουν έναν τρόπο να εκμεταλλευτούν το πιο ευνοϊκό κομμάτι της νομοθεσίας. Οπότε πρέπει να λαμβάνουμε συνεχώς πληροφορίες από τα κράτη-μέλη, γιατί όσο περισσότερα μαθαίνουμε, τόσο περισσότερο μπορούμε να ενημερώσουμε τις αστυνομίες, να τους πούμε, κοιτάξτε, έχει αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας, γιατί αυτό το οποίο ίσχυε πριν από δύο χρόνια δεν ισχύει πια. Και βλέπουμε παραδείγματος χάρη στο Ιταλικό οργανωμένο έγκλημα ε, μια μετακίνηση προς ε, δραστηριότητες χαμηλού κινδύνου. Γιατί βεβαίω αυτή τη στιγμή κάποιος συλληφθεί και περάσει 20 χρόνια στη, φυλακή για λαθρεμπόριο ναρκωτικών, άμα αποφυλακιστεί θα κάνει κάτι άλλο, έτσι δεν θα στραφεί πλέον στα ναρκωτικά. Αυτό βλέπουμε αυτή τη στιγμή, ελπίζω να απάντησα στην ερώτησή σας. Αυτό που είναι σημαντικό για να είμαστε επιτυχείς είναι να αλλάξουμε. Η Ευρωπαϊκή Αστυνομία ξεκίνησε ήδη. Πρέπει να αλλάξουμε προσέγγιση. Διευκρινίζοντας το ποινικό αδίκημα, ακινηθούμε από το να δούμε στοιχεία, να καταλάβουμε σαν επιχείρηση, να αντιληφθούμε σαν επιχειρήσεις σε αυτές οι εγκληματικές οργανώσεις. Δηλαδή, από την αρχή να μην ερευνούμε τα εγκλήματα που έχουν διαπράξει και μόνο, αλλά πώς λειτουργούν, τις οικονομικές ροές. Δεν είμαστε σε θέση να πούμε που βρίσκονται τα χρήματα και είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα. Δεν μπορούμε να είμαστε επιτυχείς αν δεν το γνωρίζουμε αυτό. Η Ευρωπόλ είναι οργανισμός εντός του οποίου μπορούμε να το κάνουμε αυτό, αν συλλέξουμε τις πληροφορίες. Κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί μόνο του να πετύχει, διότι η επένδυση σε μια χώρα, η έρευνα σε μια χώρα μπορεί να πετύχει ε, αν δεν υπάρχουν σφαιρικές πληροφορίες. Το νέο αυτό focal point προσπαθεί να συλλέξει τις πληροφορίες, να τις αναλύσει και να κάνει ανάλυση και να βοηθά τους ερευνητές των κρατών μελών ούτως ώστε να μπορούν να καταλάβουν ε, την εμβέλεια της ομάδας και συντονισμένα να την αντιμετωπίσουν. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Είναι αλλαγή προσέγγισης. Ευχαριστώ. Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, θέλω να ευχαριστήσω τη αυτή περιπτώση τους εκπροσώπους Ευρωπόλ, τον Μισελ Ρόσεμπαχ. Συνάδελφε Μάκιντάρ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς λυπούμε, διότι καθυστέρησα, ήταν απόφευκτο, δυστυχώς, και δεν μπόρεσα να ακούσω όλα όσα υπόθηκαν σήμερα το πρωί. Από αυτά που άκουσα και από αυτά που διάβασα κατάλαβα ότι το θέμα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όταν μιλούσατε για την φύση του οργανωμένου εγκλήματο στη μεγάλη επιχείρηση. Τον πιάσαν τον καπόνε για φοροδιαφυγή και όχι τίποτα άλλο. Αυτό θυμήθηκα. Ο δρόμος που ακολουθείτε είναι σωστός. Αυτό που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα ήταν ε, το έγκλημα που αφορά τα όπλα και τις πληροφορίες από τα όπλα, ε, βαλιστικές πληροφορίες ε, για να αντιμετωπιστεί το έγκλημα και να διασυνδέονται άτομα μεταξύ τους, ομάδες μεταξύ τους. Μπορείτε να μας πείτε κάποια πράγματα. Χρησιμοποίησατε πληροφορίες από βαλιστικές μελέτες για την εξυχνίαση εγκλημάτων. Τι καταφέρατε να πετύχετε όσον αφορά την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος χρησιμοποιώντας αυτή την προσέγγιση. Απάντηση. Οι δραστηριότητες Ευρωπόλ αντικατοπτρίζουν τις προτεραιότητες. Τα πιο επίγοντα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κρατημένη σε αυτό το οργανωμένο έγκλημα και τρομοκρατία δεν εστιαστήκαμε πολύ όσον αφορά το έγκλημα το σχετικό με τα όπλα. Όμως οι νέες προτεραιότητες όσοι έχουν αποφασιστεί από το Συμβούλιο Ιστορικού και Δικαιοσύνη τον Ιούνιο αναφέρουν και το εμπόριο πυροβόλων όπλων. Ήδη ξεκινήσαμε την προετοιμασία μας για να ξεκινήσουμε επιχειρησιακό πρόγραμμα όσον αφορά το εμπόριο πυροβόλων όπλων και εντός αυτής της προτεραιότητας σίγουρα ως προβλέπεται και στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα δημιουργήσουμε σχέδια δράσης, στατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια δράσης που θα πρέπει να υλοποιηθούν και εντός των σχεδίων δράσεως πιθανότατα θα έχουμε και ένα κομμάτι για ιατροδικαστικές ε, ε, αναλύσεις και την ανάλυση των βα, βαλιστικές των όπλων κλπ. Αυτά θα τα διευκρινίσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κάτι μέλη. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει τελικά. Ε, αλλά νομίζω ότι ίσως αυτό που αναφέρατε να είναι ένα ενδιαφέρον θέμα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, όπως έλεγα, θέλω να σας ευχαριστήσω για το ότι ήρθατε, για τη δουλειά που κάνατε. Ευχαριστώ τον Μισελ Ρόσεμπαχ και τον Ντάβιντ Έλερο που μας έδωσαν σήμερα και άλλες ε, πληροφορίες, ε, κάποια στοιχεία για την τελική εικόνα. Θέλουμε να διαβάσετε τις ευχαριστίες και στον ε, Διευθυντή, τον κύριο Wainwright. Υποστηρίζει η Επιτροπή αυτού του είδους τις εργασίες, αυτές τις δραστηριότητες και ελπίζουμε και στο μέλλον το επόμενο νομενό κοινοβούλιο ε, να ξέρει, να βλέπει μακριά και να συνειδητοποιήσει τη σημασία της δουλειάς σας και να δώσει συνέχεια στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ολοκληρώνουμε. 9 Σεπτεμβρίου στο Στρασβούργο η επόμενη συνεδρίαση από τις 19 μέχρι τις 20 και 30. Η γραμματεία θα σας κοινοποιήσει την αίθουσα. Θέλω να σας ευχηθώ καλές διακοπές, καλή ξεκούραση και να τα ξαναπούμε εδώ πιο αποφασιστικοί και κυρίως πιο ισχυροί ε, ούτως ώστε να μπορούμε να υποστηρίξουμε τα επιχειρήματά μας στην Ολομέλεια του Στασβούρου. Περιμένω όλους εκεί στην Σύνοδο του Οκτωβρίου